Buenas tardes. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών σήμερα, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Θα προεδρεύσω εγώ ε, για καμιά ωρίτσα μέχρι να έρθει η πρόεδρο Σεσίλια Βίκστρομ με την πτήση της. Να εγκρίνουμε καταρχά την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνεται. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Κατόπιν, να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Δεν έχει πρακτικά όμως, Επομένω δεν έχουμε σημείο 2. Και ανακοινώσεις ε, της Προέδρου επίσης δεν έχουμε. Περνάμε λοιπόν ούτε και διάφορα έχουμε και περνάμε στην αναφορά 58 2015 από την πλατφόρμα Πασχόντων από υπατήτη ΔΑΣΕ για τη δημιουργία ενός ε, ευρωπαϊκού ε, πλαισίου για την εκρίζωση της υπατήτηδας. Είναι εδώ οι αναφέροντες, ο ε, δόκτωρ Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Αγγίλιο, υπατολόγος, ο οποίος εκπροσωπεί την πλατφόρμα των ε, Πασχόντων για την υπατήτη ΔΑΣΕ ε, να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του εδώ. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον ε, ε, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Αγκούγιο. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, απευθύνομαι σε εσά εκπροσωπώντας την πλατφόρμα των ασθενών υπατήτηδας σε στην Ισπανία. Αναφερόμαστε σε ασθενείς γιατί ε, αυτά τα ε, ε, μάλλον σε πληγέντες, γιατί αυτοί οι οποίοι ε, πλήττονται από την υπατότητα ΔΑΣΕ δεν είναι μόνο οι πάσχοντες αλλά και οι συγγενείς τους. Επομένως έχουμε 56 εκατομμύρια Ευρωπαίους οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες αυτές της ασθένειας. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, πολύ υψηλότερο του συνολικού πληθυσμού της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίε και κύριοι, αυτό είναι το πραγματικό μέγεθο του προβλήματο. Το άρθρο 158 που λέει ότι ε, κατά την εκτέλεση των πολιτικών και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της υπατήτηδας στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Σε μια μελέτη του 2014 για την υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται ότι ε, από το 2013 έως το 2030, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα, οι θάνατοι από κύρωση του έπατος θα αυξηθούν από κατά 110% ε, και οι θάνατοι από υπατικές νόσους ε, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε διότι πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες θεραπεύουν μέχρι και το 95% των περιπτώσεων μια ασθένεια η οποία ήταν σχεδόν ανίατη ε, και θανατηφόρα τα τελευταία 30 χρόνια. Το σχέδιο εκρίζωσης της υπατήτηδας ΣΕ. Ε, που προτείνει η πλατφόρμα μας ε, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει στρατηγικός ε, σχεδιασμός πλήρης. Καταρχάς, ζητάμε θεραπεία για όλους, διότι μέχρι τώρα έχει πανερμηνευθεί η κατευθυντήρια γραμμή που δίνεται για τους ασθενείς. Ε, και λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς και όχι την επιστημονική πραγματικότητα ε, θεραπεύεται η μειοψηφία, ε, δηλαδή μόνο οι πολύ σοβαρές περιπτώσεις και αυτό σημαίνει ότι δεν επιλύουμε το πρόβλημα αλλά δεν αποφεύγουμε και τις δαπάνες διότι όταν κάποιος πάσει κύρωση του ύπατος θα πρέπει οι ασθενείς να κάνουν περιοδικές ε, επισκέψεις και το ίδιο ισχύει και με την ε, μέτρια χρόνια υπατήτη δασέ. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει θεραπεία για όλους τους ασθενείς με κατάλληλη περιοδικότητα. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γίνεται διάγνωση μόνο στο 25% των περιπτώσεων υπατήτη δασέ. Κατά το, σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία είναι πολύ ε, καλά καθορισμένες οι ομάδες ε, στόχος όπου πρέπει να γίνεται ε, τεστ για να εντοπιστεί ασθένεια. Επίσης υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και άλλες μολύνσεις, επομένως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κοινό πρωτόκολλο πρόληψης της ασθένειας για να ε, ε, γνωστοποιηθεί και στον πληθυσμό αλλά και στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας ε, το πρωτόκολλο και τι πρέπει να κάνουν για την περίπτωση πρόληψης της ασθένειας. Σε μία έκθεση του 2013 του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη των Νόσων αναγνωρίζεται ότι είναι επισφαλή και ανακριβή τα στοιχεία για όσους, για μολύνονται. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το HCV σε κάθε χώρα μέλος ε, και ε, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις περιπτώσεις της θεραπείας και τι συνέπειες έχει η θεραπεία για κάθε περίπτωση. Πρέπει επίσης να γίνει κατάλληλος έλεγχος ε, της ιατρικής δαπάνης. Το υψηλό κόστος των φαρμακευτικών ε, σκευασμάτων σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ακριβή η θεραπεία. Επομένως πρέπει να υπάρχουν συντονισμένοι μηχανισμοί όπως για παράδειγμα νομοθεσία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που επιτρέπει ε, να ε, διατίθενται δημόσια κάποια φάρμακα, καθώς επίσης κάποιες υποχρεωτικές άδειες για φάρμακα για θεραπεία. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένων φαρμάκων. Ο ειδικό απεσταλμένο ε, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ε, λέει ότι πρέπει να γίνει μια ε, παγκόσμια επαναδιαπραγμάτευση για την πρόσβαση σε φάρμακα όταν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μια παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. Επίσης πρέπει να διαθέσουμε ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μα για να επιλύσουμε μια βασική αντίφαση που υπάρχει μεταξύ των διεθνών συμβάσεων περί διανοητικού ίση ε, ιδιοκτησία και ε, των ε, συμβάσεων που υπάρχουν για την πρόσβαση στην υγεία. Ε, κυρίες και κύριοι, εσείς έχετε τη δυνατότητα να επιλύσετε αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι, πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε την πλατφόρμα και τον δόκτωρα Χωσελοής γιατί τόσο σαφή και ευεριστατωμένη παρουσίαση. Έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο εκπροσώπους. Η Μπελίνα Πεντολόφσκα είναι η πρώτη και στη συνέχεια ο Αλφόνσο Κάλλης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που έθεσαν αυτό το θέμα αλλά να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συμβολή του στη συζήτηση γιατί η, η ογενής υπατήτηδα γενικότερα και συγκεκριμένα η υπατήτηδα γάμα αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σιωπηλό δολοφόνος και ένα από αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τη βγάλουμε από τη σιωπή και να τεθεί πραγματικά το πρόβλημα. Την περασμένη εβδομάδα ε, δεν ήμασταν πολύ μακριά στη βιβλιοθήκη Σολβέ υπήρξε μια σύνοδος για την υπατήτητα γάμα που οργανώθηκε από ε, πολλές ε, οργανώσεις, από πολλών επιπέδων οργανώσεις και ακριβώς αυτό τονίστηκε ότι όπως είπε και ο αναφέρον πρέπει οπωσδήποτε να ε, μιλήσουμε δυνατότερα για την συγκεκριμένη ασθένεια. Συμφωνούμε λοιπόν σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπατε. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί είναι το επίπεδο δοκιμών και παρακολούθησης αλλά και βεβαίως η πρόσβαση στη θεραπεία που έχει να κάνει με ε, το ε, κατά πόσο ε, υπάρχει πρόσβαση και είναι οικονομικές, οικονομικώς ανεκτές οι τιμές. Θα ήθελα να επανέλθω πάντως στη βασική αρχή της δικής μας αρμοδιότητας. Αναφερθήκατε το άρθρο 186, 168, όμως το τελευταίο τμήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέει μάλιστα ότι η ευθύνη για τον ε, καθορισμό της πολιτικής για την υγεία, την οργάνωση και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένων ε, των ιατρικών ε, πόρων επαφίεται στα κράτη-μέλη. Επομένως όλα αυτά τα οποία αναφέρατε δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δεν έχουμε δηλαδή αρμοδιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε επίπεδο κοινοτικό, όμως μπορούμε να μην παραμένουμε αδρανείς και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν την ασθένεια αυτή. Και τι εννοώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει θεραπεία ούτε να ε, δημοσιεύσει κλινικές κατευθυντήριες γραμμές, αυτός δεν είναι ο ρόλος μας. Ε, δεν μπορούμε να πούμε στα κράτη-μέλη σε ποιες ομάδες να δώσουν προτεραιότητα και τι φάρμακα να χρησιμοποιήσουν, αλλά αυτό που μπορούμε και ήδη κάνουμε είναι υπό το πρόγραμμα υγείας να, ε, να υποστηρίξουμε την όλη προσπάθεια. Έχουμε ήδη αρκετά ε, προγράμματα που έχουν ξεκινήσει. Πέρσι μάλιστα έχουμε μια κοινή δράση που έχει δρομολογηθεί ε, ξέρετε ότι οι περισσότεροι πάσχοντες είναι χρήστες ε, ενδοφλεβίων ναρκωτικών, οπότε αυτό αποτελεί ένα από τους στόχους μας και υπάρχει και ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο διαπραγματευόμαστε για την ώρα που έχει να κάνει με την έγκαιρη, διάγνωση της υπατήτηδας. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι είναι σιωπηρός δολοφόνος, γιατί ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει κανείς την ασθένεια αυτή Υπάρχει ένα πρόγραμμα λοιπόν για το 2016 που είναι στα τελευταία στάδια έγκρισης του Αυτά είναι, ένα, αυτά είναι μερικά από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά γιατί δεν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 που είναι πολύ ευρύτερο μέσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που επενδύονται σε έρευνα υπό το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο το υπαριθμών 7 πάνω από 60 ε, ε, δισεκατομμύρια ε, δόθηκαν και τα δύο πρώτα χρόνια του ορίζοντα 2020 3,5 εκατομμύρια ευρώ ήδη έχουν δαπανηθεί σε έρευνα. Όσον αφορά τώρα την παρακολούθηση της ε, ασθένειας και την ε, επίβλεψη, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο και η το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών το έχει ήδη αναφέρει. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Τα κράτη-μέλη βέβαια έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις αναφορές τους, αλλά στις εκθέσεις τους πρέπει να αναφέρεται και για ποιο λόγο υπάρχουν ελλείψεις. Δεν ε, είναι εύκολο για μας να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτές οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών. Ε, αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Όσον αφορά τώρα τη θεραπεία και τη δυνατότητα ε, υποστήριξης, ε, το 2014 και 2015 το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία φαρμάκων ε, ενέκρινε νέα φάρμακα στα οποία νομίζω ότι αναφερθήκατε κι εσείς με την ε, επισπεσμένη διαδικασία. Προσπαθήσαμε λοιπόν όσο το δυνατόν συντομότερα να τα παρέχουμε στους ασθενείς. Άλλα μέσα ε, που έχουμε δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε άμεσα όπως σας είπα τη θεραπεία αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, υπάρχει, μια κοινή συμφωνία ε, παροχής ε, ε, που αφορά την ε, διασυνοριακή παροχή βοήθεια για τις θεραπείες, δηλαδή αν οι χώρες επιθυμούν μπορούν από κοινού να παρέχουν θεραπείες χρειάζεται, χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις ε, χώρες, πέντε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέντε ε, μέρη για να ε, ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της κοινή παροχής και έχουμε πολλές ενδείξεις από κάποια κράτη-μέλη ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Πρέπει πάντως να τονίσω ότι επαφίεται στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν μπορούμε να τους την επιβάλλουμε. Εκτός από αυτό, εμείς βεβαίως πιστεύουμε ότι όσον αφορά τις τιμές ε, και το μηχανισμό τιμολόγησης των φαρμάκων έχουν άμεση σχέση με το κατά πόσο είναι προσιτά από απόψεως τιμής ε, τα φάρμακα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και έχουμε προγράμματα και υπό το πρόγραμμα υγείας ε, αύξησης της διαφάνειας της τιμολόγησης των φαρμάκων και νομίζω ότι έχω καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα του φάσματος των ε, ε, μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένο αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, χρησιμοποιώντας το, αξιοποιώντας το για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση ε, Ανάπτυξης που είναι εδώ για να καλύψουν τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, που αναφέρατε επίσης. Θα ήθελα να συνοψίσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την υπατήτη γάμα ως ε, σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντιπαραβολή με την υπατήτη Β δεν υπάρχει και εμβόλιο για την υπατήτη Γ. Πρόκειται λοιπόν για ένα ιστορικό σε μια ιστορική χρονική στιγμή ε, ακόμη ε, και αν σκεφτούμε σε 10-15 χρόνια ότι μπορούμε να εξουδετερώσουμε την ασθένεια αυτή, πρέπει να υπάρχει θέληση να το κάνουμε. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά φάρμακα τα οποία είναι αποτελεσματικά σε μεγάλο βαθμό. Και εμείς θέλουμε να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Γενική Διεύθυνση Growth από την ε, Διεύθυνση για τις Δημόσιες ε, Συμβάσεις. Θέλω να συμπληρώσω λίγο τόσο η συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και να δούμε αν οι ψηλές τιμές των φαρμάκων συνιστούν παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. Γενικά πρώτος στόχος της δημόσιας Συμβάσεις είναι να ανοίξει η αγορά στον ανταγωνισμό για να μπορέσουν οι ε, ενδιαφερόμενοι να έχουν καλύτερες συνθήκες και να πιάνουν τόπο τα χρήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει σαφής ε, περιγραφή για το πώς προκυρήσεται ένας διαγωνισμός για μια δημόσια προμήθεια. Είναι πάρα πολύ διαδικαστικοί οι κανόνες. Δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια λοιπόν που να εξασφαλίζουν ψηλές ή χαμηλές τιμές. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο διαγωνισμό μπορούν να συνασπίζονται σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο ή και μεταξύ κρατών μελών και να κάνουν κοινή προσφορά. Και εκτός ε, της συμφωνίας, βέβαια χωρίς βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μπορείτε να λέτε ότι συγκεντρώνουμε τις ανάγκες μας και προκυρήσουμε ένα διαγωνισμό για τις προμήθειες. Και έτσι έχετε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Για μικρές χώρε, όπως είναι οι χώρες τη Βαλτικής είναι ενδιαφέρον να προκυρήσουν κοινού διαγωνισμούς για να έχουν πιο ισχυρά ε, ανταγωνιστικά επιχειρήματα και διαπραγματευτικά απέναντι στη βιομηχανία. Ε, δεν είναι κανόνας λοιπόν και μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα εάν εκείνοι που προκυρήσουν το διαγωνισμό είναι, επαναλαμβάνω, ε, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να προκυρηθεί κοινό διαγωνισμό για εκδήλωση ενδιαφέροντο. Εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Αλφόνσο Κάλε. Ευχαριστώ, γεια σα. Να δω, μιλήσω ισπανικά. Σωστά ισπανικά, γιατί μου μπαίνουν και κάτι αγγλικά στη μέση. Εγώ εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Grow, ανάπτυξη δηλαδή, εσωτερική αγορά και βιομηχανία, σε μια μονάδα που ασχολείται με βιομηχανική ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς προτείνουμε την νομοθεσία, την εκπονούμε, το νομοπαρασκευαστικό ε, στάδιο για ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία, στο Ευρωπαϊκό Σήμα κτλ. Οπότε, ένα από τα θέματα που μας απασχολούν είναι οι φαρμακευτικές ευρεσιτεχνίες και η προστασία αντίστοιχη της πνευματικής ιδιοκτησίας των φαρμακευτικών εταιριών. Τα όσα είπαν οι συνάδελφοι με καλύπτουν απολύτω και είναι πολύ εύστοχα για να μην μακρηγορώ εγώ και να βοηθήσω να προχωρήσει η συζήτηση για την υπατήτη δασέ στην ε, τοποθέτησή σας μιλήσατε και για ενδεχόμενα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στα πλαίσια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θέλω λίγο να σας εξηγήσω πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Λοιπόν, όλα αυτά τα φάρμακα τέτοιου τύπου, ε, όπως αυτά της υπατίδας, ε, προστατεύονται από ευρεσιτεχνίες με αποκλειστική διάθεση στην αγορά όσο διαρκεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστατεύονται. Βεβαίως τέτοια φάρμακα είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί ε, ε, είναι τεράστιες επενδύσεις πάνω από ένα δις ευρώ για να αναπτύξεις ένα νέο φάρμακο και για, από την αρχή της έρευνας μέχρι την είσοδό του στην αγορά μπορεί να περάσει και δεκαετία. Οπότε να μπορεί μια φαρμακευτική, ένα εργαστήριο να ε, έχει αυτές τις επενδύσεις και επί μία δεκαετία να κάνει επενδύσεις και έρευνα αν δεν ξέρει τι θα γίνει, αν θα πετύχει το φάρμακο, αν θα έχει οικονομική επιτυχία. Γι' αυτό χρειάζονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Είναι ένα πολιτικό εργαλείο για να προστατεύει την έρευνα και να ενθαρρύνει. Και να ενθαρρύνει, λέγω, τι φαρμακευτικέ εταιρείε να ρισκάρουν ε, αυτά τα χρήματα και να κάνουν αυτή τη δουλειά και αυτό το εμπόριο και να κυκλοφορούν τα προϊόντα τους, τα φάρμακά τους στην αγορά καλή η στα φάρμακα και ε, σημαντική, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει το φάρμακο. Εκεί βοηθάνε οι πατέντες και τα διπλώματα ευρεσιταχνία να γίνονται καινοτομίε. Το πρώτο στάδιο είναι να βρεις το φάρμακο και μετά να το αγοράσεις και πόσο θα κάνει και να κυκλοφορεί στην αγορά. Αλλά πρέπει να εφευρεθεί το φάρμακο και να κυκλοφορήσει. και από εκεί και πέρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε νομοθετικά μέτρα για τη διευκόλυνση ε, των γενοσύμων ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπατε κι εσείς. Υπάρχει κοινοτική νομοθεσία που λέγεται Provision για τα γενώσιμα ε, που μπορούν να αναπτύσσονται από πλευρά έρευνα, καθώ ακόμα διαρκεί η ευρεσιτεχνία, για να μπορεί γρήγορα να βγει στην αγορά το γενώσιμο όταν λήξει η πατέντα. Υπάρχει μια στρατηγική για την ενιαία αγορά ε, στα τέλη του 2015 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει πώ μπορεί να διευκολύνει τα γενώσιμα και την έρευνά του για να υπάρχει μεγαλύτερη καινοτομία και μόλι λήξει η πατέντα να είναι έτοιμο το γενώσιμο να κυκλοφορεί στην αγορά. Επίση, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πριν από λίγα χρόνια έκανε κάποιε μελέτε για να δούμε πώς θα μπορούσαν να μπαίνουν πιο εύκολα στην αγορά τα γενώσιμα. Εγώ ασχολούμαι με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου εφαρμόζει κάτι που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζεται ε, συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη και στις διμερείς συμφωνίες και η δική μου γενική διεύθυνση και το δικό μου τμήμα ασχολείται με διεθνή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα διεθνή οργανισμό ε, των Ηνωμένων Εθνών που ε, ονομάζεται Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Βέβαια, το δίπλωμα βρεσιτεχνία δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλείδε και ε, εξαιρέσει. Για να μπορούν να κυκλοφορούν γρήγορα και τα γενώσιμα. Επομένω, τα αναφέρετε κι εσεί, τα γνωρίζετε σήμερα που είναι οι υποχρεωτικές άδειε. Εκτός αυτού υπάρχει και ένα θέμα ε, απαλωτρίωσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε πάρα πολλές αρμοδιότητες. Το κοινοτικό κεκτημένο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι αρκετά περιορισμένο. Οι πατέντες ρυθμίζονται από μια διεθνή συνθήκη και σύμβαση που δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η σύμβαση του Μονάχου που εκεί είναι και το γραφείο το Ευρωπαϊκό για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και από εκεί και πέρα εθνικές νομοθεσίες. Και σε ό,τι αφορά την απαλωτρίωση των δικαιωμάτων και τις υποχρεωτικές ε, άδειε κυκλοφορίας, εκεί ισχύει το εκάστοτε εθνικό δίκαιο. Το Ισπανικό δίκαιο, για παράδειγμα, για τις ευρεσιτεχνίες προβλέπει την απαλωτρίωση και την αφαίρεση δηλαδή της αποκλειστικότητας από την εταιρεία και το, θέμα των υποχρεωτικών αδειών. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Επίσης, δεν έχουμε διαπιστώσει να ζητεί κάποιος εναρμόνιση του δικαίου ευρωστητεχνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εργαζόμαστε επί των θεμάτων αυτών γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αν εσείς ασχοληθείτε με την εθνική σας νομοθεσία και προκειμένου την ισπανική, υπάρχει το άρθρο 73, το 86 καθώς επίσης και το 90 όλων αυτών των νόμων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανική κυβέρνηση θα μπορούσε να απαλωτριώσει, να αφαιρέσει δηλαδή την αποκλειστικότητα από την ε, εταιρεία που έχει την ευρεσιτεχνία και να δηλώσει ότι κυκλοφορεί υποχρεωτικά αυτό το φάρμακο στην αγορά για να αρχίσει να παράγεται. Αυτά είχα να σας πω. Σας είπα στην αρχή πώς δουλεύουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς ε, μας απασχολεί η ευρεσιτεχνία, τι σημαίνει μια πατέντα, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ενθαρρύνει ε, την ε, καινοτομία, τη φαρμακευτική δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Ε, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, μπορείς να αφαιρέσει την πατέντα, ε, μπορείς να αρχίσεις να κάνεις έρευνα για γενώσιμα όσο διαρκεί η ευρεσιτεχνία κτλ. Υπάρχουν διεθνείς διαπραγματεύσεις, διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Muchas ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα τα, ο λόγο στα μέλη. Έχουμε ένα κατάλογο, αλλά όποιος θέλει να παρέμβει μπορεί να ζητήσει το λόγο. Η κυρία Άουκεν καταρχάς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Ορισμένες φορές ε, φαίνεται ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν τα λόμπι τους και κάθονται εδώ μας λένε πως έχει κατάσταση με έναν τρόπο που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να προσφέρουμε κατάλληλη θεραπεία για αυτή την ασθένεια. Διότι πρόκειται για σαφέστατη ληστεία. Είναι ληστρική συμπεριφορά προς τον ε, δημόσιο προπολογισμό για την υγεία. Από ό,τι κατάλαβα ε, είναι είναι υψηλότερο 50.000% το φάρμακο. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία Αγγίλα το αγόρασε από άλλη εταιρεία που σημαίνει ότι δεν έχουν κόστος για έρευνα και ανάπτυξη. Έχει παρέλθει προπολού το κόστος αυτό. Και επίσης, δεν ξέρω αν οι αναφέρονται μπορούν να ενημερώσουν, υπάρχουν ε, κάποιες παρενέργειες τις οποίες γνωρίζουν πώς να θεραπεύσουν αλλά περιμένουν να θεραπεύσουν αυτές τις παρενέργειες όταν κοντεύει να εκπνεύσει σχεδόν ε, το φάρμακο για να το παρατείνουν άλλα 20 χρόνια και να επιβαρύνουν και για άλλα 20 χρόνια τον προϋπολογισμό για την υγεία. Είμαστε σε απελπισμένες περιπτώσεις όταν συζητάμε για την ανθρώπινη ζωή και ορισμένες φορές αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κανόνας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι υπάρχει αρκετή δύναμη από πλευρά μα να αντιμετωπίσουμε αυτού του μεγάλου ισχυρού τη φαρμακοβιομηχανία. Να σας πω επίσης ότι πρώτον και κυριότερον, εμείς, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, κατά πάσα πιθανότητα, εγώ είμαι από τη Δανία, δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Αλλά μαζί θα πρέπει να ζητήσουμε πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την τιμολόγηση. Προσπαθεί να γίνει αυτό στι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, όπου τα λόμπι το σταμάτησαν, αλλά χρειάζεται πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την τιμολόγηση. Γιατί τιμάται κατά αυτή την τιμή ένα φάρμακο, πόσα είναι ε, από τις ομάδες πίεσης ε, και μάρκετινγκ και ποιο από αυτό το τμήμα του, του τιμήματος είναι έρευνα και ανάπτυξη. Και επίση, ε, ε, όσον αφορά την απολωτρίωση του διπλώματο ευρεσιτεχνία, ε, το θέμα εδώ είναι ο θάνατό στη ζωή μου. Είναι θέμα επιβίωση και ορισμένοι άνθρωποι θα πεθάνουν επειδή ακριβώ ο κλάδο δεν προσαρμόζεται καθόλου σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν γνωρίζει ποια είναι η πραγματική τιμή αυτών των προϊόντων. Γνωρίζετε ποιο είναι το κόστος για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα, στη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα. Γνωρίζετε τίποτα για πιθανές παρενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να θεραπευθούν ήδη από τώρα αλλά προσπαθούν να το παρατείνουν για να ανανεώσουν το δίπλωμα ευρεσιτεχνία. δεν το ξέρω καλά αυτό το θέμα. Υπάρχουν επίσης και κανόνες TRIPS που θα μπορούσαμε ίσως να τους επικαλεστούμε ε, για το συμφέρον της ανθρώπινης υγείας. Και θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε τις τιμές στη φαρμακοβιομηχανία, διότι αυξάνονται κατακόρυφα οι τιμές και οι ασθενείς είναι τα θύματα. Ορισμένες φορές ε, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη και είναι απλώς κερδοσκοπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε πρέπει πλέον να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν θα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον. Γιατί αυτό ήταν το τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται εκεί και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σύγκρουση συμφερόντων να φύγουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά και για του άλλου οργανισμού, αλλά είναι σαφέστατο αυτό στον Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ. Gracias. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κιουτεντάλεν και αυτό Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και, στους, και τους αναφέρονται. Εγώ είμαι μέλος της ομάδας φίλων του Ήπατος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί στο, στη βορειοανατολική Αγγλία είναι τεράστιο το επίπεδο ε, θνησιμότητα λόγω της ασθένειας αυτής, κυρίως λόγω της φτώχειας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καταθλιπτικό αυτό και αν δει κανεί πώ χρησιμοποιούνται, πώ αξιοποιούνται ε, οι ιατρικοί πόροι έρευνας και ανάπτυξη. είναι πάρα πολύ λίγο αυτό το τμήμα ε, που λαμβάνει η σχετική έρευνα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι αναφέροντε είναι εδώ Ήμουν στη Σύνοδο Κορυφής που αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα και κάποιοι, υπήρξαν στοιχεία που καταδεικνύουν ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει δράση και από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι πρέπει με ε, την, με την, με την φυματίωση, με, ε, με τον ιό HIV και με την υπατήτη γάμα πρέπει να συνδέσουμε την έρευνα αυτή γιατί ακριβώς ε, αυτοί οι άνθρωποι ε, οι άνθρωποι που πάσχουν από όλες αυτές τις ασθένειες υποφέρουν τρομερά. Πάρα πολύ καλό αυτό που είπε η ε, κυρία Άουκεν. Είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει κα, και να συμπληρώσει κάποια πράγματα από αυτά που είπε γιατί τα είπε σχεδόν όλα. Πάντως κάτι άφησε ε, που μπορούμε να το πούμε και εμείς. 23 μέλη συμμετέχουν τώρα στην ε, Συμφωνία κοινή Παροχής Φαρμάκων. Το μόνο που μένει να δούμε τώρα είναι πώς θα το προωθήσουμε. Με τέτοιο τρόπο όπω να εξασφαλίσουμε ότι ε, τα, ε, ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αγορά των φαρμάκων ώστε να μειωθεί το κόστος. Όσον αφορά τώρα το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εγώ δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να, υπάρξει περισσότερη, περισσό, να υπάρξουν περισσότεροι όροι στε, για τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων ώστε ε, τα κονδύλια έρευνας να κατανοήσουν ανέμονται καλύτερα και πιο δίκαια και αυτό το είπε και η κυρία Άουκεν σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το τελευταίο που είπε όσον αφορά ε, το τέλος της, ε, του, της ευρεσιτεχνίας. Περιμένουμε δηλαδή να φτάσουμε στο τέλος την εκπνοή της ευρεσιτεχνίας για να την ανανεώσουμε. Νομίζω ότι σε σχέση με αυτό το evergreening της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει οπωσδήποτε να το ξαναεξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα την ε, δυνατότητα αξιολόγησης από τη δυνατότητα δικτύων αξιολόγηση τεχνολογίας ώστε να συνάδει περισσότερο με το άρθρο, ε, της, το άρθρο 15 της οδηγίας 24 ε, του 2011 όσον αφορά την αξιολόγηση της τεχνολογίας για να μπορέσουμε να ε, βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην αξιολόγηση της έρευνάς τους Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω, ε, να πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολείται κυρίως με τα θέματα των μεταδοτικών ασθενειών ε, και οι συνάδελφοι από τους Βρετανούς εργατικούς που είναι επίσης μέλη της ομάδας φίλων του Ήπατος θα ήθελα να πω ότι μπορεί εντός της Επιτροπής Περιβάλλοντος να υπάρξει προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό και θα ήθελα να προτείνω ειδικότερα μια προφορική ερώτηση που θα συνδέει την υπατήτη δαγάμα με το σχέδιο δράσης για τον ε, HIV όπως ε, ε επίσης ε, και η, σχέση των, η σχέση μεταξύ των τριών αυτών ιών που ανέφερα προηγουμένως. Και αυτό πρέπει να συνδεθεί με ε, το αίτημα η οδηγία ε, περί διαφάνειας ε, να ενημερωθεί και αυτό να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με το από πού προέρχονται αυτές οι υψηλές τιμές και να μην παραμένουμε εχμάλωτοι όμοιροι των φαρμακευτικών βιομηχανιών για φάρμακα τα οποία χρειάζομαστε σε, κατεπηγόντως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια επιδημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Eh. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους της πλατφόρμας των πληγέντων και των ασθενών. Ένα χρόνο μετά τη συνάντησή μας επιτέλους έρχονται να καταθέσουν την αναφορά τους προσωπικά και θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια του έτους αλλά και προηγουμένως από τότε που η πατήτηδα σε κυριάρχησε στην ισπανική επικαιρότητα έγινε πρώτη είδηση Πέρασαν πολλές μέρες, πέρασαν πολλοί μήνες. Και ποια είναι η διαφορά ε, με τις μέρες που περνούν ε, για να έρθει μια αναφορά ή μια άλλη. Εδώ μιλάμε για ζωές ανθρώπινες και κάθε μέρα που περνάει μπορεί να χάνονται ζωές. Και αυτή είναι η διαφορά με τις υπόλοιπες αναφορές. Το θέμα δεν είναι μόνο να λύνουμε τα προβλήματα που φθέτουν υπόψη μας οι πολίτες, αλλά πρόκειται για τη ζωή τους. Να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε είναι μια χρόνια ανίατη θανατηφόρα ασθένεια στο παρελθόν, η οποία σήμερα ε, μπορεί να ιαθεί. Και θα πρέπει ε, να αντιδράσουν αντίστοιχα με την ίδια ευθύνη οι πολιτική. Μας έφερε αντιμέτωπου με του εαυτού μα είπατε τη Δασέ, μα έβαλε ένα καθρέφτη και μα έδειξε ότι δεν λειτουργεί. Κάτι πάει στραβά στην κατάσταση με τα φάρμακα. Θα πρέπει να ανασκουμποθούμε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το ξέρω ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, η τιμολόγηση και η ε, οικονομία της δημόσιας υγείας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και η εντολή της αυτή να εγγυάται την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θυμάμαι την τελευταία συνεδρίαση στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια με ειδική συζήτηση για την πρόσβαση στα φάρμακα. Και σύμφωνα και με την αναφορά αυτή θέλω να πω ότι θα πρέπει η Κομισιόν και το Συμβούλιο επιγόντως να καταρτήσουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο πρόσβασης στα φάρμακα που να περιλαμβάνει πολλά από τόσα λέμε εδώ. Εγώ δεν θέλω να ποινικοποιήσω ούτε τι φαρμακευτικέ ούτε τα λόπη, ούτε τι κυβερνήσει, ούτε κανέναν. Ο καθένα τη δουλειά του κάνει και η δουλειά η δικιά μας πια είναι να συνεργαστούμε όλοι για ένα κοινό στόχο. Το σχέδιο αυτό, το ευρωπαϊκό, θα πρέπει να προβλέπει μια νέα σχέση με την φαρμακοβιομηχανία, γιατί είναι απαραίτητη η εταίρη μα για την εγγύηση της δημόσιας υγείας, που δεν χωρά καμία αφιβολία γι' αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί η οδηγία για τη διαφάνεια στην τιμολόγηση των φαρμάκων, να δούμε εκβάθρον ξανά το θέμα της ευρυσιτεχνίας. να μην συνδέεται το κόστος της έρευνας με το τελικό κόστος στην τιμή του φαρμάκου. Δηλαδή, θα υπολογίζουμε πόσο έχουμε επενδύσει στην έρευνα και θα το χρεώνουμε στον τελικό ασθενή. Και θα πρέπει τα κράτη να εξασφαλίζουν βασικά φάρμακα για τους πολίτες. Σήμερα έχουμε τους ενδιαφερομένους, τους πληγέντες που αγωνίζονται για τη ζωή τους και για τη ζωή των αγαπημένων τους για να έχουν ένα δικαίωμα να τους δοθεί μια θεραπεία που υπάρχει ήδη. Και είναι δική μας εντολή να το κάνουμε αυτό. Να εξασφαλίσουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εγώ απλώς θα ήθελα τώρα να ε, προτείνω το εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το σκεφτούμε. Στην Ευρώπη καταφέραμε να βάλουμε ένα φραγμό στην περιαγωγή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα φάρμακα και να σώσουμε ζωές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπατρίς. Θα προσπαθήσουμε λίγο να περιορίσουμε το χρόνο, διότι έλεγε και η Πρόεδρος ότι πρέπει να δώσουμε και τη δυνατότητα σε αναφέροντα από άλλα σημεία να μιλήσουν. Επομένως, ε, τρία λεπτά από εδώ και πέρα σε όποιον λάβει το λόγο. Ο κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν είχα επιλογή το πότε θα πάρω το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο από του προαλήσαντες συναδέλφου, και να σας πω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δίλημα. Επί τη ουσίας ε, συμφωνώ με το σύνολο σχεδόν των επιχειρημάτων που ακούστηκαν και από τους αναφέροντες ε, ένα μεγάλο τμήμα των όσων υπόθηκαν από τους προλαλήσαντες παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην ανήκουμε στην ίδια πολιτική ομάδα. Παρ' όλα αυτά είμαστε η Επιτροπή Αναφορών και δεν είμαστε εδώ ε, για να συζητάμε απλώς και να φύγουμε όλοι από εδώ και να μην έχει προχωρήσει το θέμα καθόλου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να επιφέρει κρίση όσον αφορά την ουσία, απλώς μπορούμε να δούμε κατά πόσο αυτή η διαδικασία η οποία ισχύει αυτή τη στιγμή μπορεί να καρποφορήσει ή όχι. Εμείς ε, πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων και η εφαρμογή από εκτελεστικής απόθεως ενός προγράμματος υγείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι εντός των, ε, εντός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τώρα, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που είναι το εκτελεστικό στέλεχος ε, δεν θέλει από μόνη της να ξεκινήσει μια πολιτική υγείας κοινή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την επιβάλλει στα κράτη-μέλη τότε είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε γιατί ε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν για να λύσουν το πρόβλημα και βλέπουμε το κουράγιο αυτών των ανθρώπων ε, που με τα ε, που έκανα το ταξίδι ε, ως εδώ σήμερα, ναι, πράγματι ε, υπάρχει δυνατότητα να, προχωρήσουν, ε, να προχωρήσει το πράγμα. Ε, το να λέμε εμεί εδώ ότι ναι, θα επιβάλλουμε σε κάθε ένα από τα 28 κράτη της Ένωσης να αλλάξουν ε, τις συνθήκες για να υπάρξει μια κοινή ενιαία πολιτική υγείας, αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Αν λοιπόν αυτό θέλουμε να επιτύχουμε, εγώ θα έλεγα να κλείσουμε την αναφορά αυτή να την παραπέψουμε στι αρμόδιε. Ε, επιτροπές και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν άλλες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως για παράδειγμα μια προφορική ερώτηση κοινή από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, ε, και ώστε να είναι ακόμη πιο ευρία η απήχηση από ότι στο πλαίσιο μιας ε, απλής Επιτροπής Αναφορών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα ως προς τις αρμοδιότητες αυτές τις οποίες δεν έχουμε για την ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μαριάς. Μικρόφωνο σα. Μικρόφωνο κύριε Μαριά. Καταρχά, να συγχαρώ του αναφέροντε που πήραν αυτή την πρωτοβουλία και ήρθαν να θέσουν αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα ε, διότι η πατήτηδα σε πράγματι είναι μια επικίνδυνη ασθένεια σε ορισμένες χώρες έχει πλήξει πάρα πολλούς πολίτες και θα έλεγα ότι εν ώψη και των μεγάλων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που παρουσιάζονται μπορεί να έχουμε και επιπλέον επιδημία της ε, ασθένειας αυτής. Άρα λοιπόν το θέμα είναι σοβαρό. Το δεύτερο είναι ότι από τη συζήτηση αναδείχθηκαν ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε το θέμα αυτό. Διότι βεβαίως ε, οι πολιτικές δημόσιας υγείας ανήκουν στα κράτη-μέλη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος κανόνας αφορά το ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική άσκηση της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων εταιριών. Και αυτό το προβλέπει η ίδια η συνθήκη. Όταν μια εταιρεία έχει μια ισχυρή θέση μέσα στην αγορά και την αποκτά αυτή την ισχυρή θέση λόγω της έρευνας που κάνει, λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων, λόγω της πατέντας και καταχράτε τη δημόσια θέση που έχει, την ισχυρή αυτή θέση, Έχουμε παραβίαση της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως έχουμε αρμοδιότητα εμείς και κυρίως η Κομισιόν να ελέγξει κατά πόσο οι συγκεκριμένες εταιρείε που κρατούν αυτή την πατέντα και την τιμολογούν με ένα αυξημένο τρόπο που να εκμεταλλεύονται επί της ουσίας τους ίδιους τους ασθενείς παραβιάζουν τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Και εγώ νομίζω ότι έχουμε μια κλασική παραβίαση διατάξεων περί ανταγωνισμού το οποίο πρέπει να το δούμε. Το επόμενο θέμα είναι η πρόσβαση των ασθενών ε, στα φάρμακα. Κάτι που το συζητήσαμε ε, στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Διότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα. Επιπλέον, εδώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μέσα στο Horizon 2020 που είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, επομένως έχουμε αρμοδιότητα εμείς ως Επιτροπή να το συζητήσουμε και να το εξετάσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε μια σειρά θέματα που νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να κλείσει η υπόθεση, πρέπει να την αφήσουμε ανοιχτή, πρέπει να δούμε τι άλλα μέτρα θα πάρουμε. Δεν είναι θέμα δικό μας επιβάλλουμε μια πολιτική στα κράτη-μέλη, αλλά δικό μας θέμα είναι πώς οι αναφέροντες που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν πρόσβαση στα φάρμακα, θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο φάρμακο και θα μπορούν οι ίδιοι να στηρίξουν τους συγγενείς τους και οι ίδιοι να πάρουν αυτά τα φάρμακα για τη σωτηρία της υγείας τους. Και γι' αυτό πρέπει κατά τη γνώμη μου να μείνει ανοιχτή υπόθεση και συγχαίρω ξανά τους αναφέροντες για την πρωτοβουλία της και την παρουσία τους εδώ. Gracias. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς <laughs> να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν γνωρίζω καμία τροποποίηση της συνθήκης για να γίνει συντονισμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φυματίωση, την ελονοσία και το HCV. Παίζουμε ουσιαστικά με τις λέξεις εδώ και λέμε ότι πρέπει να αλλάξει συνθήκη. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η ρήτρα για την προστασία που έχει κάποιους περιορισμούς, διότι ε, ο καθορισμός της τιμής και το πώς παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε όμως πολλές δυνατότητες και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι λίγο πιο αυστηρή. Δεν ζητάει κανένας χρήματα, λογικό δεν ζητάμε χρήματα, αλλά σίγουρα είναι πολύ ακριβή έρευνα. Θα ήθελα όμως να μου δώσετε αυτά τα στοιχεία για να γνωρίσουμε ακριβώ ποια είναι τα στοιχεία για την έρευνα από πλευράς ε, της φαρμακοβιομηχανίας. Επίση, θυμάμαι ότι υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αμφισβητεί τα στοιχεία που μα δίνουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Όχι ότι καταφέρουμε κατά των φαρμακοβιονοχωνών, αλλά νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση συμπεριφέροντων μεταξύ πνευματική ιδιοκτησία που περιέχει ε, τη δυνατότητα 20 χρονών μονοπωλίου ε, και το θέμα είναι όμω ότι η προστασία τη υγεία είναι κάτι τελείω διαφορετικό, είναι τελείω διαφορετικό αγαθό και δεν θα πρέπει να τα ε, συσχετίσουμε αυτά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνία τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ρόλο να διαδραματίσει καταρχά ω προ του πολίτε. Διότι ξέρουμε ότι το 25% των ανθρώπων που γνωρίζουμε ότι έχουν, ε, είναι ασθενείς πατήτηδα ΣΕ, μα λείπει το υπόλοιπο 75%, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιο εδώ στην αίθουσα που να πάσχει από πατήτηδα ΣΕ και να μην έχει διαγνωστεί. Επίση, πρόκειται για μια ασθένεια που αυτή τη στιγμή μπορεί να θεραπευτεί και υπάρχουν πάρα πολλοί σημαντικές συνέπειες γιατί ε, λείπει ένα μόνο μέτρο να προσπαθήσουμε να εκριζώσουμε αυτήν την ασθένεια. Και νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που είναι αυτά που πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε, να τους δώσουμε μια ανάλυση και πώς να βρουν μια ισορροπία με αυτό το σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς μπορούν να βρουν τα θέματα τη έρευνα ε, των φαρμάκων. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς από εδώ να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαφάνεια, για την τιμολόγηση των φαρμάκων, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει. Επίσης, από τον ορίζοντα 2020 θα μπορούσαμε να ζητήσουμε δημόσια χρηματοδότηση έρευνας και αυτά τα χρήματα τα οποία επέτρεψε να, δημιουργήσει, να μια νέα καινοτομία, να μην ε, μπορεί να τα εκμεταλλευτεί μόνο η φαρμακοβιομηχανία. Επομένω, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να γίνουν. Θα ήθελα λοιπόν ολοκληρώνοντα να ευχαριστήσω και να ζητήσω το εξή. Να ευχαριστήσω την πλατφόρμα για την υπατήτη ΔΑΣΕ που ανέβασε του τόνου. Διότι ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσες μεγάλες αποκλήσει ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίνει μάχη είναι γιατί πραγματικά αυξήθηκαν οι τόνοι σε αυτή τη συζήτηση και γίνεται μια πραγματική συζήτηση και σας ευχαριστούμε που το κάνατε αυτά γιατί αύριο θα είναι οι ασθενείς ε, που πάσουν από καρκίνο ή οι ασθενεί από άλλε ασθένειε. πρέπει να του προσφέρουμε τι κατάλληλε λύσει από πλευρά Ευρώπη από τι δυνατότητε που έχουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνοντα να σα πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Και επομένω γι' αυτό και το θέμα θα έπρεπε να συζητηθεί στην Ολομέλεια, να γίνει μια προφορική ερώτηση και να δούμε πώ μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα συντονισμένο σχέδιο από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκρίζωση τη υπατήτηδα ΣΕ. Για αυτού του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν, να το μάθουν και να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα ώστε να θεραπεύονται οι ασθενεί. Τίποτα άλλο ευχαριστώ. χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την πλατφόρμα των πληγέντων από την Υπατήτη σε μια ασθενής και το περιβάλλον τους για τον αγώνα τους που πραγματικά είναι ένα αγώνας υπερπάντων και υπερόλων. γιατί κάποια στιγμή μπορεί ο καθένας από εμά ανά πάσα στιγμή να προσβηθεί από υπατήτητα σε. Όπως είπαν και αναφέροντες, υπάρχουν φράγματα ε, που αυξάνουν τις ε, πιθανότητες μέχρι 95% να ιαθεί η πατήτητα σε. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το φάρμακο όμως, στον κόσμο συνεχίζει κάθε μέρα να πεθαίνει κόσμος εκατοντάδε κάθε χρόνο από υπατήτητα σε. Και στην ίδια την Ευρώπη συνεχίζουν να πεθαίνουν. Και για ποιο λόγο, διότι πολλές κυβερνήσεις δεν επιδοτούν τη θεραπεία. Οπότε στο Ισπανικό κράτος η κυβέρνηση δεν επιδοτεί τα φάρμακα για όλους και το Ισπανικό κράτος μπορεί να δει ένα κόστος 25.000 ευρώ για 12 ε, εβδομάδες. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, έχουν ευθύνη και οι κυβερνήσεις που δεν επιδοτούν τη θεραπεία, αλλά θα πρέπει να στοχεύουμε πολύ πιο ψηλά στις μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Γιατί γι' αυτό φταίνε αυτοί που είναι αστρονομικές οι τιμές, οι πατέντες προστατεύουν τα κέρδη των φαρμακευτικών εταιριών. Δεν χρειάζονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, όπως είπε πρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι θανατική καταδίκη οι πατέντες για εκατομμύρια κόσμου. Για να βγάζουν λεφτά φαρμακευτικές εταιρείες και να σωρεύουν κέρδη και μηδενικά ε, στο τραπεζικό τους λογαριασμό. 13,3 δις δολάρια έβγαλε μια εταιρεία, ε, ε, αυτή που παράγει το Σομπάλτι. Και θα πρέπει να συζητάμε άλλα πράγματα τώρα για έρευνα, δημόσια, για δημόσιες φαρμακευτικές βιομηχανίες που να μπορούν να δίνουν όλα αυτά τα φάρμακα. Είναι γεγονός ότι η αρμοδιότητα για τη δημόσια υγεία είναι των κρατών μελών, αλλά επίσης είναι γεγονός, και εκεί είναι βασικά το πρόβλημα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητες για τις ευρεσιτεχνίες. Και αυτό είναι το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να ενδιαφέρεται και να ανταποκρίνεται περισσότερο για τα συμφέροντα των μεγάλων φαρμακευτικών πολυεθνικών εταιριών παρά για τους πολίτες άνδρες και γυναίκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιπλέον αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται το TTIP. Μην το ξεχνάει αυτό κανείς. Και πιέζουν οι μεγάλες φαρμακευτικές για να μπουν ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να ενισχυθούν και να εμποδιστούν τα γενώσιμα. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να απαιτήσουμε. Να σταματήσει ε, το TTIP ε, να υποκλίνεται στη συμφέροντα των μεγάλων φαρμακευτικών. Και έρχονται εδώ διάφοροι βουλευτές και λένε μεγάλα λόγια και μετά ψηφίζουν υπέρ του TTIP. Λίγη στοιχειώδης συνέπεια χρειάζεται. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει στην Ολομέλεια να κάνουμε προφορική ερώτηση για να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται και τι βήματα κάνει και τι μέτρα λαμβάνει για να εξασφαλίσει ότι θα έχουν θεραπεία όλοι οι πολίτες που τη χρειάζονται. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τι προτίθεται να κάνει ή τι θα έπρεπε να κάνει για να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία πάντα για τα διπλώματα εύρεση τεχνίας. Τελειώνω. Σήμερα επίση, μετά τη συζήτηση αυτή και τις διάφορες παρεμβάσεις φάνηκε σαφώς ότι αυτό που ψάχνει η Ευρωπαϊκή ε, διαμεσολαβήτρια για τις ε, σχέσεις που υπάρχουν ε, και τη διαπλοκή μεταξύ εργαζομένων σε μεγάλες σε διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι κάτι που θα έχει συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο αναφέρον έχει τον λόγο τώρα για δύο-τρία λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ. Ε, <clears throat> σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας όλους και θα ήθελα να σας προτρέψω αυτή τη φορά να μην ξεχάσετε τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της επατήτηδας C. Την πρώτη φορά που εγκρίθηκε δήλωση για την επατήτηδα C στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν στις 29 Μαρτίου του 2007. Είμαστε στο 2016 πλέον, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωράμε τόσο αργά, δεν μπορούμε να είμαστε ανέστητοι ενώπιον τόσο σοβαρών προβλημάτων όπως κατέστησα θες ότι αυτό είναι. Επιπλέον, θα ήθελα να σχολιάσω ότι είναι προφανές ότι η έρευνα πρέπει να έχει και ένα όφελος. Δεν μπορεί να είναι ένα όφελος, ένα κέρδος το οποίο θα στερεί ε, τα μέσα από τα κράτη-μέλη να θεραπεύσουν τους ασθενούς τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω τώρα που αλλάζουν ε, οι συνθήκες, πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες για τις ε, διεθνείς συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί επηρεάζουν τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που ε, έχουμε σχέση ο ένας με τον άλλον και αυτό είναι θεμελιώδη σημασία. Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαι με τη θεραπεία της υπατήτηδας και πλέον ο ορίζοντας της ελπίδας δεν πρέπει να απογοητεύει ούτε τους πολιτικούς, ούτε τους εκπροσώπους, ούτε κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς, λοιπόν. Θα κάνω την εξή πρόταση και θα, μου πείτε τη γνώμη σας. Από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι συνάδελφοι ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και με βάση την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στείλουμε μια επιστολή προς την ε, ε, τον Επίτροπο τον Αρμόδιο, τον κύριο Ανδρουικάητης, για τη δημόσια υγεία και τα τρόφιμα, να πούμε τι διεμήφθη εδώ, να δούμε τη δική του άποψη και επίσης να στείλουμε μια επιστολή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή που λέγεται ΕΝΒΗ και είναι αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, να δούμε τι θα μας πει και εκείνη και μετά θα κάνω την πρόταση να στείλουμε επιστολή και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας διότι προετοιμάζεται τώρα την πρώτη παγκόσμια στρατηγική για την ιογενή υπατήτηδα και καλό θα ήταν να δούμε και αυτό το παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα την προφορική ερώτηση που ζητήσατε για την Ολομέλεια, καλό θα ήταν να περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής και του Επιτρόπου και να το συζητήσουν οι συντονιστές για να αποφασίσουν εκεί, όχι στο Ολομέλεια της Επιτροπής. Δεν το αποκλείω, αλλά να περάσει από τους συντονιστές πρώτα. Πώς τα βλέπετε. Η Σολεδά τη ζήτησε πρώτο λόγο. Η προφορική ερώτηση για μένα είναι απαραίτητη. Και η, μόνη αναβολή που δέχομαι είναι ε, ε, να κάνει η ΕΝΒΗ, η αρμόδια επί της ουσίας και η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, ε, να έχει μία πρωτοβουλία για την Ολομέλεια. Και μην μου λέτε να απαντήσει ο Επίτροπος, γιατί να περιμένουμε την απάντηση του Επιτρόπου. Αυτή η απάντηση δεν με ικανοποιεί καθόλου. Μόνο αν κάνει κάτι η ΕΝΒΗ θα δεχτώ αναβολή της προφορικής ερώτησης. Αν δεν αναλάβει καμία πρωτοβουλία η ΕΝΒΗ, τότε η δική μας επιτροπή να το κάνει. Αν το κάνει η ΕΝΒΗ, μαζί. Η κοινοβουλευτική θα πρέπει να είναι η πρωτοβουλία, όχι να περιμένουμε απαντήσει κομισιών. Εάν συμφωνείτε, να το κάνουμε έτσι. Η ΕΝΒΗ ε, ε, ε, επιστολή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιστολή, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Επιστολή και να δούμε τι θα μας απαντήσει η ένβη για να κάνουμε την προφορική ερώτηση. Συμφωνείτε να κλείσει η κυρία Άουκεν. Απλώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ακριβεί στι ερωτήσει που, κάνουμε, που θέτουμε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν να του ζητήσουμε το εξή. Για το συγκεκριμένο προϊόν να υπάρξει διαφάνεια όσον αφορά την τιμολόγηση. Η ιστορία αυτού του προϊόντος, του φαρμάκου, φάνηκε ότι δεν αφορά καθόλου την έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι πολύ συγκεκριμένη η περίπτωση αυτή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στην ερώτησή μας ως προς την υπατήτηδα γάμα. Και νομίζω ότι η τιμολόγηση το ιστορικό της όλης διαδικασίας και να ρωτήσουμε τι διαδικασίες μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κράτη-μέλη των οποίων ε, η θέση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο ε, αν έπρεπε να ακολουθήσουν την λογική των φαρμακοβιομηχανιών 50.000% της τιμής δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι σε ερωτήσεις μας, να φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη στρατηγική και όχι να πλατιάζουμε προς όλες κατευθύνσεις. Από ό,τι κατάλαβα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ως προς αυτήν την πολύ, τις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, μια ερώτηση που περιλαμβάνει και όλες τις ανησυχίες ε, της κυρίας Σάουκεν. Ε, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης και να δώσω τώρα το λόγο στην Πρόεδρο, η οποία θα αναλάβει και την Προεδρία της συνεδρίας από εδώ και πέρα. Thank you so much and thanks to... Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι εδώ στην πρώτη αυτή ε, συνάντηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε και ε, θα ήθελα να περάσω και στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης ευθύς αμέσως που είναι το υπαριθμόν 6 και είναι η αναφορά που αφορά την κατασκευή ενός κέντρου σιδεροδρομικών τεχνολογιών στη Μάλαγα της Ισπανίας Νομίζω η κυρία Αλβιόλ εκπροσωπεί ε, τον αναφέροντα και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο ευθύς αμέσως. Oh, Παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα για να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάτασης. Κυρία Αλβιόλ. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο συζητήθηκε κάποια στιγμή. Ε, φαίνεται ότι δεν ε, ζητήθηκε χρηματοδότηση για το σχέδιο αυτό, αλλά ε, επομένως θεωρώ ότι μάλλον θα μπορούσε να κλείσει η αναφορά. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αν κάποια στιγμή η Ισπανική κυβέρνηση ξαναυποβάλει το σχετικό σχέδιο ή υπάρξει κάποια σχετική πρόταση, θα πρέπει να ξανανοίξει η αναφορά χωρίς να πρέπει να ε, ξαναπεράσουν οι αναφέροντες από όλη τη διαδικασία και να ξανανοίξει με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί, εάν και εφόσον ξανακατατεθεί το σχέδιο. Μάλιστα πάρα πολύ σύντομη η εισαγωγή σα στην αναφορά αυτή. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά ονόματα έχω εδώ μπροστά μου. Ο κύριο Ράμο Φλωρίδο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, στο σημείο αυτό θα συζητήσουμε μαζί δύο αναφορές την 240 το 2011 και τη 1536 το 2012 και επειδή το θέμα αφορά διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα παρέμβουν ε, εκπρόσωποι από τρεις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα θα μιλήσω εγώ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιβάλλοντος θα σας συνοψίσω λίγο την πρόταση και θα σας εξηγήσω τι έγινε από περιβαλλοντική σκοπιά και μετά θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής ε, και Αστικής Πολιτικής για να σας ε, αναφέρει τα περί πιθανής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και τέλος στο συνάδελφο Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τις πτυχές που σχετίζονται με την ε, πιθανή κρατική επιχορήγηση για τα θέματα αυτά. Όπως σας είπα, πρόκειται για δύο διαφορετικές αναφορές που εκπροσωπούν δύο διαφορετικέ οργανώσει, οι οποίε όμω θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν τον ίδιο στόχο, διότι αφορούν το λεγόμενο πρόγραμμα εγκαταστάσεις δοκιμής ε, για το Κέντρο Τεχνολογίας της Αντεκέρα στην ε, περιοχή της Μάλαγα, στην αυτόνομη περιοχή της Ανδαλουσίας ε, στην Ισπανία. Πρόκειται για το σιδηροδρομικό δακτύλιο της Αντεκέρα, έτσι είναι γνωστό το πρόγραμμα πρόκειται για την παραγωγή ενός ε, μεγάλου κυκλώματος ε, δοκιμών ε, για τροχαίο υλικό και, σιδη, και σιδηροδρόμους ταχείας κίνησης και έχουμε την περιοχή της Μάλαγα, την Αντεκέρα και τη Φόντεντε Πιέδρα που θα ε, περιλαμβάνει η περιοχή. Υπάρχει η δημόσια επιχείρηση Άντις ε, που ανήκει στο Υπουργείο Χωροταξίας της Ισπανίας ε, η οποία θα είναι αρμόδια για την κατασκευή του έργου. Οι αναφέροντες είναι αντίθετοι στο σχετικό έργο για τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν όσον αφορά την καταστροφή του περιβάλλοντος καθώς επίσης και το γεγονός ότι επειδή πρόκειται για μια περιοχή η οποία έχει μεγάλο γεωργικό πλούτο και επίσης είναι αντίθετοι για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ζητούν να επιλεγεί μια άλλη περιοχή για αυτό το ε, ε, σχέδιο δοκιμών ε, σιδηροδρόμων. Στην ε, μία από αυτές τις αναφορές ε, ζητήθηκε να εξεταστεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς ξεκινήσαμε μια επίσημη έρευνα και αποτανθήκαμε στις Ισπανικές Αρχές ζητώντας πληροφορίες για το σχέδιο αυτό, το σχετικό έργο και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών οδηγιών που θα έπρεπε να εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση, την ε, οδηγία για τις περιβαλλοντι... μελέτη περιβαλλοντικών υποπτέσεων, την οδηγία Natura 2000 και την οδηγία για τα πουλιά υπήρξε μια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ισπανικών Αρχών και τα τελευταία χρόνια λάβαμε απαντήσεις από το Υπουργείο Χωροταξίας, ε, από την εταιρεία την κατασκευαστική την Άντις, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από την ε, Ανδαλουσία. Και επίσης Πρέπει να πω ότι από περιβαλλοντική σκοπιάς ε, υπήρχε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκριση του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε με μία δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων τον Νοέμβριο του 2011 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα ε, της 24ης Νοεμβρίου του 2011. Επίσης, οι Ισπανικές Αρχές ισχυρίζονται ότι δεν ε, αφορά την οδηγία Natura 2000, διότι η περιοχή η οποία επελέγει έχει αποφύγει περιοχές ε, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσε ε, από πλευρά οικοτόπων. Επομένως, δεν αφορά η σχετική οδηγία. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες ε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ε, ε, πληροφορίες για το κατά πόσον θα υπάρξει, θα υλοποιηθεί το έργο. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, λοιπόν έκλεισε την έρευνα γιατί δεν μπορεί να είναι ανοιχτή επαόριστον και θα πρέπει επίσης να σας πω τέλος ότι ε, υπήρξαν αρκετές προσφυγές στα εθνικά δικαστήρια από τις διάφορες οργανώσεις και πλατφόρμες οι οποίες αντιτίθενται στο έργο αυτό ε, και σε διοικητικά και σε ποινικά δικαστήρια και σε κάποιες, κάποιες από αυτές τις προσφυγές εκκρεμούν ακόμα και τα εθνικά δικαστήρια μπορεί να γνωρίζουν και κάποια πράγματα που να αφορούν ε, θέματα πέραν της εφαρμογής των οδηγιών που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά λοιπόν από τη δική μου παρουσίαση για το περιβάλλον να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής να σας πει τα περί πιθανής χρηματοδότησης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο του σχετικού έργου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο απευθεία ε, στο συνάδελφό σας και μετά τον εκπρόσωπο της ε, γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού. Για να σας έχουμε ακούσει και τους τρεις, παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν συντομότεροι, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Πολιτική Αστική. Να σας ενημερώσω για αυτό το μεγάλο έργο ε, από τα Διαστατικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι ένα μεγάλο έργο. Έχει ζητηθεί κοινοτική χρηματοδότηση πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο κατέθεσε η Ισπανία επέβαλε την υποψηφιότητα το Δεκέμβριο του 2011 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για τα τεχνολογικά και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τις παρατηρήσεις της το Μάιο του 2012 στην πρόταση αυτή. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος ήταν τακτικές οι επαφές με τους ε, κοινωνικούς εταίρους και φορείς που ήταν αντίθετοι, περιβαλλοντικοί φορείς, περιφερειακοί και μια πλατφόρμα ε, που ήταν αντίθετη με ε, την κατασκευή και επίσης οργανώσεις γροτών. Έκαναν ερωτήσεις κοινοβουλευτικές, αναφορές και άλλες διαμαρτυρίες. Η Ισπανία μετά τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τη τεχνική, οικονομική και άλλη σκοπιμότητα και περιβαλλοντική απάντησε μέρη στις παρατηρήσεις αυτές και κάποια στιγμή επειδή δεν απάντησε σε όλες, σκέφτηκε να αποσύρει αυτό το μεγάλο έργο και τον Ιούλιο του 2013 να καταθέσει νέα εκδοχή της πρότασης αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε παρατηρήσεις, η Ισπανία δεν απαντούσε σε όλες τις παρατηρήσεις και το έργο δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί όπως λέγει ο κανονισμός εντός μιας περίοδου μέχρι το 2017 ε, και η Ισπανία αποφάσισε να αποσύρει αυτό το μεγάλο έργο από την κοινοτική χρηματοδότηση. Οπότε το ΕΣΠΑ που τρέχει 13-17 δεν μπορεί να καλύψει ε, το πρόγραμμα, ούτε πρόκειται στη συνέχεια μέχρι το 17 να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Um, um... Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι εδώ εκπροσωπώντας την ε, Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού και θα ήθελα να σας δώσω λίγο περισσότερες ε, λεπτομέρειες οι Ισπανικές ε, αρχές ενημερώνουν ενημέρωσαν ε, ε, τις δημόσιες αρχές χρηματοδότησης και κρατικής ενίσχυσης το 2012 και κάνοντας το αυτό είπαν ότι το κάνουν μόνο για, νόμους, για λόγους ασφάλειας δικαίου γιατί θεωρούν ότι ολόκληρη δημόσια ε, χρηματοδότηση των 358 εκατομμυρίων ευρώ που καλύπτεται πλήρως από τον Ισπανικό προϋπολογισμό και το ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, ε, θα μπορούσε να ισχύει μόνο, κατά πόσο, μόνο στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί συγχρηματοδότηση και χρηματοδότηση από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μόνο στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης. Το Μάρτιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη διαδικασία ερευνών ε, για το θέμα αυτό και το έκανε γιατί ακριβώς ε, διαπίστωσε ότι σε αντίθεση με την άποψη των Ισπανικών αρχών αυτή η χρηματοδότηση θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση και δεν θα συν δεν θα συμμορφωνόταν με τους ε, κανόνες ε, περί έρευνας ε, και ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις αμφιβολίες της λέγοντας ότι δεν είναι απαραίτητη γιατί υπήρχε περίπτωση ε, κατάρρευσης ολόκληρου του ε, σχεδίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο υπήρχαν αποδιστικά στοιχεία ε, για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δοκιμών. Και θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε όντως λόγος αν δεν είχαν ληφθεί υπόψη κανενός είδους ιδιωτικές επενδύσεις. Και υπήρχαν αμφιβολίες επίσης από πλευράς μας ότι στο πλαίσιο του RNDI ε, οι σχετικοί κανόνες δεν έγιναν σεβαστοί. Σε αυτή την επίσημη λοιπόν διαδικασία έρευνας η οποία έχει ήδη ξεκινήσει οι Ισπανικές αρχές ε, και οι και φορείς εμπλεκόμενοι ε, φορείς της αγοράς ε, συμμετείχαν σε σχέση με ε, τους ενδεχόμενους ανταγωνιστές αυτών των εγκαταστάσεων δοκιμών και ε, όπως ε, ανέφερα, η έρευνα αυτή ε, έχει δρομολογηθεί, εξακολουθεί να υφίσταται και γίνεται ανάλυση αυτή τη στιγμή των αποτελεσμάτων που λαμβάνουμε, της πληροφόρησης που έχουμε λάβει κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης των ερευνών μας και ελπίζουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια απόφαση μέχρι την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στους Ευρωβουλευτές. Κυρία Αλβιόλ, θα έχετε ε, βεβαίως το λόγο στο τέλος ε, της ε, του θέματος αυτού, επειδή ούτως ή άλλως μιλήσατε ως εκπρόσωπος ε, του αναφέροντος. Ξέρετε ότι ο δεύτερος αναφέρον δεν είναι παρόν, οπότε θα πρέπει να τη συζητήσουμε μαζί, θα λάβετε το λόγο στο τέλος. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Όχι, άρα κυρία Ερβιόλ έχετε το λόγο. Ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ σύντομα. Ιδού ένα παράδειγμα για το πώς ο γόνας ο κοινωνικός πιάνει τόπο. Καμιά φορά αυτός ο σιδηροδρομικός δακτύλιος ρίμαζε το περιβάλλον, τη γεωργία και το σύμπαν εκεί πέρα. Και χάρη στην πλατφόρμα, όχι στο δακτύλιο, ε, εγκαταλείφθηκε το έργο και χάρη στη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αυτή η έρευνα και πραγματικά θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Καμιά φορά οι κοινωνικοί αγώνες αποδίδουν ε, πιάνουν τόπο και αποφέρουν κάπως. Να κλείσει η αναφορά γιατί δεν έχει ζητηθεί χρηματοδότηση μέχρι την περίοδο αυτή. Αν κάποια στιγμή επανέλθει η πρόταση θα το ξαναπούμε, να ξανανοίξει η αναφορά. Ευχαριστώ. Και ο γόνα τώρα δικαιώνεται. Mm-hmm. Η κυρία Καμπεσόν θέλετε και εσείς το λόγο. Ναι, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι πράγματι το έργο είναι ένα έργο, μα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα περί χρηματοδότηση, ε, που θα έχει σημαντικά οικονομικά ωφέλη για την περιοχή. Μα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι από πλευρά περιβαλλοντική δεν υπάρχει καμία παραβίαση τη οδηγία. Επομένω, ε, ε, τα περιβαλλοντικά προφυλάσσονται τουλάχιστον. Επομένω, το πρόβλημα είναι ότι είναι πρόβλημα χρηματοδότηση. τι γίνεται με την πηγή χρηματοδότηση και πόσο συνάδει αυτό με τα κονδύλια τα οποία θα δοθούν. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν το ενδιαφέρον που υπάρχει από πολιτική σκοπιά από την κυβέρνηση και δεν ε, ε, έψεξε κανείς κάποια εναλλακτική λύση. Ε, τώρα, το κατά πόσο θα πρέπει να κλείσουμε ή όχι την αναφορά. Ε, εάν την κλείσουμε και αν ξανανοίξει, αν ξαναυποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση, μπορούμε να το συζητήσουμε όταν θα το ξανασυζητήσουμε. Ω προ την ασυμβατότητα των κονδυλίων και των ταμείων. Εάν υπάρχει τέτοια συμβατότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσει ότι πρέπει να συζητηθεί, τότε αυτά θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και τότε θα πρέπει ε, να γίνει τη χρηματοδότηση βάσει των όσων προβλέπονται και από τα ταμεία. Ευχαριστώ. Ωραία. Κάνουμε μια ισπανοϊσπανική συζήτηση τελικώς. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ναι, κοιτάξτε η αναφορά αυτή δεν ήταν μόνο για τη χρηματοδότηση, ήταν για πολλά θέματα και διάφορα, όπως το ζήτημα ότι κάποιοι δήμοι θα ήταν ε, ε, έγκλειστοι εκεί ένας θύλακος, ε, μέσα στο δακτύλιο, θα υπήρχαν προβλήματα για τη γεωργία, για το περιβάλλον γενικά. Δεν είναι μόνο χρηματοδότηση. Αν ξανάρθει το έργο για να ζητήσει χρηματοδότηση, θα πρέπει να ξανανοίξει αναφορά όπως έχει κατατεθεί και για τα υπόλοιπα θέματα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Okay, fine. Ε- Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και προηγουμένως, δύο είναι οι αναφορές, είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Ε, η δεύτερη εστιάζει περισσότερο στο, στην πτυχή του ανταγωνισμού και η πρώτη αναφορά ε, την, τον αναφέροντα του, της οποίας εκπροσωπείτε εσείς αφορά περισσότερο το περιβαλλοντικό κομμάτι. Πρέπει πάντως ε, να πω ότι αυτό δείχνει θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει μια Επιτροπή Αναφορών ότι έχει ε, μια άποψη και μπορεί να διαφωτίζει τέτοιου είδους υποθέσεις θέσεις υπό διάφορες ε, οπτικές ε, γωνίες και απόψεις. Όπως και η κυρία Αλβιόλ ε, μας είπε, εμεί κάναμε τη δουλειά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνη συνεχίζει τη δουλειά της εν προκειμένου. Μπορούμε πάντως να κλείσουμε και τις δύο αναφορές. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, αυτό έχω σκοπό να κάνω. Ευχαριστώ πολύ, μπορούμε να προχωρήσουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η γνωμοδότηση για τη διασυνοριακή αναγνώριση των υιοθεσιών. Και όπως γνωρίζετε, το Μάιο η Επιτροπή μας όρισε εισηγητή τον κύριο Μαριά ε, ως συντάκτη γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θέλαμε να, ε, ε διαφωτίσουμε τα ε, σημεία ε, της πρότασης που λάβαμε, όπως επίσης ε, και τα αποτελέσματα μιας εξεταστικής των πραγμάτων επίσκεψης στο Λονδίνο πέρυσι, που ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική και χρήσιμη επίσκεψη. Τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης ε, θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες πολύ σύντομα σε όλους τους συναδέλφους. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει διάσταση απόψεων, οπότε δίνω το λόγο σε εσά κύριε Μαριά σύντομα και ε, μετά στους υπολείπους συναδέλφους. Παρακαλώ να είμαστε σύντομοι όμως γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία που είχαμε για αυτή την ε, γνωμοδότηση όπως επίσης και τη γραμματεία της Επιτροπής γιατί πράγματι συνέβαλε στο να διαμορφώσουμε μια γνωμοδότηση η οποία έχει γενική αποδοχή θα έλεγα. Το θέμα της διασυνοριακής αναγνώρισης των υιοθεσιών είναι πολύ σημαντικό. Έχει απασχολήσει με σειρά αναφορών που έχουν γίνει στην Επιτροπή μας. Μια διάσταση ε, επίσης ε, έχει να κάνει με τις υιοθεσίε οι οποίες ε, ε, είναι αναγκαστικές, δηλαδή χωρίς την συγκατάθεση των φυσικών γονέων ε, και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Επομένως το πρώτο που θίγουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι είναι ότι αυτό που πρέπει να πριτανεύει κάθε φορά σε κάθε απόφαση για την ε, διακρατική αναγνώριση των υιοθεσιών είναι το συμφέρον του παιδιού, το συμφέρον του τέκνου, διότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια δικαίου για να γνωρίζουμε τι ισχύει σε κάθε κατάσταση. Να προστατεύονται τα δικαιώματα των γονέων και των παιδιών και να τηρούνται φυσικά οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως οι διατάξεις που έχουν σχέση με την ηθαγένεια. Διότι θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια αποτελεί τη βάση από την οποία πηγάζουν συγκεκριμένα δικαιώματα και για τους γονείς και για τα τέκνα διότι όλοι έχουν στην περίπτωση που είναι πολίτες βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών έχουν και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Το τρίτο θέμα είναι να αποφεύγουμε τις υπερβολικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις ενώ το επόμενο στοιχείο που πρέπει να μας απασχολεί είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιζήμιες συνέπειες οι οποίες υπάρχουν για υιοθεσίες χωρίς τη συγκατάθεση των φυσικών γονέων και των ε, θετών παιδιών. Νομίζω αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το έχουμε συζητήσει και πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολήσει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τους κανονισμούς, τον κανονισμό 2203-01 του 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά να, έχουμε, ε, να εξετάσουμε και άλλες πλευρές όπως είναι η, σε περίπτωση υιοθεσία να μπορούν οι συγγενείς των φυσικών γονέων να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη μόνιμη φροντίδα του παιδιού. Νομίζω ότι αυτά είναι κυρία Πρόεδρε τα βασικά σημεία της ε, γνωμοδότησης αρκετά σύντομα και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, να ακούσουμε και τους συναδέλφους και να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now the floor... Ευχαριστώ πολύ και τώρα η Κυρία Πιτέρα πρώτη. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σύμβαση της Χάγης διέπει τις διεθνείς υιοθεσίες και μετά έχουμε την αυτόματη αναγνώριση. Ε, Συνεπώ, υπάρχει ασφάλεια δικαίου εν προκειμένου. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σε σχέση με τις εθνικές νομοθεσίες και την αναγνώριση αυτών μεταξύ των κρατών μελών όταν έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο υιοθεσία και μετά οι γονείς αποφασίζουν να ε, μετακομίσουν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση, αναγνώριση και το, οι Βρυξέλλες 2 δεν αναγνωρίζουν, δεν, δεν το ρυθμίζουν αυτό. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Να σα πω ένα παράδειγμα. Οι γονείς αποφασίζουν ε, να μετακομίσουν σε ένα άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το γύψη λόγο. Εκείνοι αποφασίζουν όμως στη χώρα στην οποία θέλουν να μετακομίσουν δεν αναγνωρίζεται η οθεσία τότε η οικογένεια δεν μπορεί να λάβει επιδόματα τέκνων, δεν μπορεί να εγγράψει το παιδί ε, στο Δήμο στον οποίο διαμένει, να το εγγράψει σε σχολείο, δεν μπορεί να έχει ατροφαρμακευτική περίθαλψη ε, και κάλυψη για το παιδί αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικοί κανόνες ε, ε, των κρατών μελών της Ένωση σε σχέση με τις υιοθεσίε. Για παράδειγμα, τα ηλικιακά όρια είναι διαφορετικά στην Ιταλία από ό,τι στην Πολωνία. Επίσης, ο ορισμός της, ε, του τι είναι οικογένεια μπορεί να διαφέρει. Κάποια κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ως οικογένειες ε, ε ομοφιλοφιλικά ζευγάρια. Σε άλλες χώρες ε, μόνο τα έτεροφιλοφιλικά ζευγάρια θεωρούνται οικογένειες. Υπάρχουν επίσης και διαφορετικοί κανόνες σε σχέση με το ποια παιδιά μπορούν να ε, υιοθετηθούν. Ε, οι κανόνες σε σχέση με το κατά πόσο πρέπει να, πώς πρέπει να γίνεται η συγκατάθεση των βιολογικών γονέων. Σε άλλε χώρε μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο, σε άλλε χώρε δεν μπορεί. Ε, οπότε νομίζω ότι ο εισηγητή δεν έχει απαντήσει στο βασικό ερώτημα. Χρειαζόμαστε την αυτόματη αναγνώριση οθεσίας εντό Ευρωπαϊκή Ένωσης και αν ναι, τι είδου ε, αναγνώριση πρέπει να είναι αυτή. Ιδάλω, ε, πώ θα λύσουμε το πρόβλημα. Θεωρεί ο εισηγητή ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνε ε, ε αναγνώριση. Α, μάλιστα. Αυτά είναι ερωτήματα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Καμπεσόν. Ε, εκ μέρου του κυρίου Κοζολίνο, του συναδέλφου μα, που δυστυχώ δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, εκπροσωπώ τον κύριο Κωστολίνο. ό Πολύ λίγα θα πω, γιατί αλλιώ θα χάσω και εγώ τη σειρά μου. Να σας πω τι μου ζητάει συνάδελφος να πω. Λοιπόν, πρέπει να εγγυάται πάντα αυτό το οποίο πρέπει να προέχει είναι το συμφέρον του ανηλίκου κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας και αυτή η αρχή η οποία φαίνεται ζωτική σημασία αλλά δεν γίνεται πάντα σεβαστή. Επίσης ζητά βάσει του άρθρου 21 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη το 1989 να ε, τεθούν σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχει διακίνηση παιδιών και να αποφύγουμε αυτή τη διακίνηση η οποία όπως είδαμε ακόμα και με την κρίση των προσφύγων ότι εξακολουθεί να είναι μια τρομακτική πραγματικότητα. Επίσης ζητά αμοιβαία αναγνώριση των αρχών και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο το ισιοθεσίας ε, βάσει τη σύμβασης της Χάβης, Χάγης του 1993 και ζητά να υπάρχει ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις ισιοθεσίες και να αποφύγω αποφεύγονται, αποφεύγονται ε, θέματα όπως ε, οι ε, διαφορές περί δικαστηρίου και φυσικά οποιαδήποτε αγοραπολισία παιδιών. Επίσης, σε περίπτωση διεθνούς υιοθεσία, όταν υπάρχει κάποιο διεθνές στοιχείο στην υιοθεσία, θα πρέπει να ενημερώνονται και να συμμετέχουν όλα τα μέρη τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία και επίσης ε, να ακούγεται και η άποψη του παιδιού σε όλη τη ε, διάρκεια της διαδικασίας και να γίνονται βάση της πρόσφατης νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σε περίπτωση διαφορών ε, ε, να πρέπει να προέχει το συμφέρον ε, του παιδιού και ε, να προστατεύεται επίσης και το συμφέρον των βιολογικών γονέων. Επίσης, εγώ από πλευρά μου να πω ότι σε αυτή τη γνωμοδότηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική πραγματικότητα τη σήμερον ημέρα. Γίνονται πολλαπλές υιοθεσίε και υπάρχουν διάφορα είδη ζευγαριών και θα πρέπει να αναγνωρίζονται κάθε ε, διαφορετικό είδο ζεύγους που θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί και να προσαρμοστούμε στην κοινωνική πραγματικότητα του σήμερα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελεονόρα, θέλεις να πάρεις το λόγο ως ε, συντονίστρια της ε, ομάδας σου. Ναι, ευχαριστώ. Η κυρία Εύη. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι πρέπει να οριοθετήσουμε το πεδίο δράσης μας. Από τη μια έχουμε τα νομοθετικά στοιχεία που είναι όλα όσα αφορούν ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία την οποία σαφέστατα πρέπει να γνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς και όπου μπορούμε να παρέμβουμε προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση ε, κυρίως όσον αφορά την ευημερία του παιδιού, ε, θα πρέπει να το κάνουμε. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλα μέσα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά την ευωμερία του παιδιού και κυρίως αυτή την περίπτωση και την αναγνώριση της υιοθεσία που αφορούν τη λεγόμενη ήπια νομοθεσία, το soft law, τα μη νομοθετικά ε, στοιχεία, τα οποία όμως πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το Κοινοβούλιο μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ συμφωνώ σε πολλά με τα όσα έχει γράψει ήδη ο συντάκτης της νομοδότησης και ήθελα απλώ να προσθέσω κάποιες ε, σκέψεις. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη αυτόματης αναγνώρισης ε, της υιοθεσία, ώστε να υπάρχει και εναρμόνιση του θεσμού αυτού στην Ευρώπη, διότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά επίσης θα πρέπει να μπορούμε να επισέλθουμε και λίγο περισσότερο στις λεπτομέρειες ε, των πρακτικών αυτών, ώστε να κατανοήσουμε και με βάση τις αναφορές που έχουμε λάβει και την Εξεταστική Επιτροπή που κάναμε ε, το γεγονό ότι πρέπει να λάβουμε πάρα πολλέ ε, πτυχέ υπόψη. Παραδείγματο χάρη, την υποστήριξη προ την οικογένεια, κυρίως προ του γονεί, που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, και θεωρούνται ακατάλληλοι γονείς. Ε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να μπορούμε να ζητήσουμε από τα ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά αρμόδια όργανα να υποστηρίξουν έστω και με οικονομική στήριξη ε, τους γονείς ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ως γονείς. Θα πρέπει δηλαδή να ε, συνδράμουμε στην ανοικοδόμηση της οικογένειας ώστε να μπορέσουν οι γονείς αυτοί να φροντίσουν ε, τα παιδιά τους. Επίσης, κάτι ακόμα όσον αφορά την ε, έννοια ότι προέχει το συμφέρον του παιδιού. Το έχουμε επικαλεστεί επανειλημμένως. Ε, δεν υπάρχει σαφής ορισμός ε, και ενιαίος ορισμός. Υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευέλικτος και αφήνει περιθώρια ερμηνεών και με βάση πολιτιστικές αναφορές και διάφορες χώρες καταγωγής. Επομένως είναι απαραίτητο να εξετάσουμε όσο το δυνατόν βαθύτερα το θέμα για να καθορίσουμε σαφώς ε, τι εννοούμε με τον όρο το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να πω αφορά όχι μόνο την ανάγκη να εναρμονίσουμε το θεσμό της υιοθεσίας αλλά να εμβαθύνουμε και σε κάποιες πρακτικές che riguardano gli affidi, affidi che σε θέματα που αφορούν ε, προσωρινή κυδαιμονία. Ε, χάνεται πολλές φορές αυτός ο προσωρινός χαρακτήρας και γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις μόνη υιοθεσία όλη αυτή η διαδικασία. Ε, η προσωρινή επιμέλεια χάνεται και γίνεται μόνιμη διαδικασία. Ορισμένες φορές έχουμε κάποιες υποχρεωτικές υιοθεσίες, υιοθεσίες οι οποίες γίνονται χωρίς τη συνένεση των ε, ε, βιολογικών γονέων. Ε, στην περίπτωση της επίσκεψης που κάναμε στη Μεγάλη Βρετανία είδαμε κάποια περιστατικά, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά και σε άλλες χώρες μέλη. Κατά την άποψή μου λοιπόν πρέπει να εμβαθύνουμε και στο σημείο αυτό και να μην παραμείνει χωρίς ορισμό και το θέμα αυτό που ε, πλήττει πάρα πολλούς γονείς ε, στην Ευρώπη με βάση και τις αναφορές που λαμβάνουν. Thank you, Ευχαριστώ, Ελεονόρα. Και τώρα, ο Εντουάχ Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, θα πρέπει να υπάρχει συνενετική εδώ αντίληψη, αλλά επειδή αλλάζουν τα ήθη και εξελίσσονται, θα πρέπει εμείς να προβλέψουμε μελλοντικές αναφορές που τυχόν μας έρθουν εδώ. Έχω μια υπόθεση που θα ήθελα να σας υποβάλω. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το συζητήσουμε για να βοηθήσουμε τους μέλλοντες γονείς. Και ε, αυτό είναι η με παρένθετες μητέρες. Σε πολλές χώρες αυτό ε, είναι αφισβητήσιμο, γίνονται πολλές συζητήσεις, πολύ οξίες, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ε, νομικό κενό. Γιατί σε κάποιες χώρες ακόμα και το παιδί αφισβητείται, η ύπαρξή του δεν αναγνωρίζεται. Είναι ένας τύπος υιοθεσίας, βεβαίως διαφορετικός από αυτόν που έχουμε συνηθίσει, αλλά ε, η κοίηση για τρίτο με παρένθετη μητέρα είναι κάτι που ε, μπορεί να γίνει αύριο νόμος κάποιου κράτους, γιατί αλλάζουν και οι νόμοι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά μπορεί να είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό να το κρίνω. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους μέλλοντες γονείς να καταλάβουν τι γίνεται και εάν και κατά πόσο μπορούν και εκείνοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Διότι, για να είμαι ειλικρινή, σήμερα ποιο είναι το καθεστώ ενό παιδιού που γεννιέται μετά από κύση ή από παρένθετη μητέρα. Εδώ σα θέλω, ξέρει κανεί να μου πει, ε, είναι νομικό κενό, γίνονται πολλέ συζητήσει με τεταμένα πνεύματα και με πάθο, αλλά ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω, το θέτω στην κρίση σα, αλλά το υποβάλλω στη συζήτηση και στο φίλο εισηγητή. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς ε, νεύει ε, καταφατικά ό,τι κάνουμε εμείς θα είναι προς το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πάντα που είναι ακριβώς ταυτόχρονα πάρα πολύ ακριβές και πάρα πολύ ασαφές όπως η όλη συζήτηση. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι είναι γνωμοδότηση αυτή. Ο κύριος Μαριάς δεν πρόκειται να γράψει βιβλίο για το θέμα αυτό αλλά μια γνωμοδότηση απλή Οπότε να μην παραφορτώνουμε τη βάρκα. Επίσης συμφωνήσαμε να συστήσουμε και μια ομάδα εργασίας για θέματα ευημερίας των παιδιών. Θα πρέπει λοιπόν να μένουμε στην ουσία, δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να προτείνει τίποτα. Να προσθέσει μάλλον, όχι, δεν τι να προσθέσει, η γνωμοδότηση είναι, τι να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρω το λόγο, αλλά έχουμε ένα παρόμοιο θέμα να συζητήσουμε αύριο, οπότε θα δω κατά πόσο αύριο θα λάβουμε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να σας ε, πω ότι είστε ευπρόσδεκτοι βεβαίως στην αυριανή μας ε, συζήτηση. Κάθε πράγμα στον καιρό του όμως, ε, ακόμα και αυτή η συζήτηση. Να δούμε τώρα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο. Μα ήμουν πάρα πολύ σύντομο στην εισαγωγή μου και θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα των συναδέλφων. Συμφωνήσω με την ε, κυρία Καμπεθόν ε, για την παρατήρηση που έκανε για την διακίνηση των παιδιών. Σε αυτή τη φάση έχουμε πάρα πολλά παιδιά που κινούνται στο πλαίσιο των τεράστιων προσφυγικών ροών τα είδαμε αυτά τα παιδιά, είχα επισκεφθεί και την Σάμο και τη Λέσβο και την Ιδωμένη ε, στα σύνορα με τα Σκόπια και είδα ότι υπήρχαν πολλά παιδιά ασυνόδευτα. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Βεβαίως συμφωνώ με την παρατήρησή σας ότι εδώ μιλάμε για μία γνωμοδότηση. Δεν συντάσσουμε την έκθεση. Η έκθεση συντάσσεται από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Επομένως αυτή έχει τη βασική ευθύνη. Το δεύτερο θέμα που τέθηκε από τη συνάδελφο του ΕΠΠ Έθεσα ένα θέμα σε σχέση με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε και να έχουμε ε, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ορισμένα προβλήματα. Τα προβλήματα αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Άκουσα τα παραδείγματα που έφερε η συνάδελφος από το ΕΠΠ που ήταν σκιώδης εισηγήτρια ότι υπάρχει περίπτωση κάποιοι πολίτες που πάνε σε άλλο κράτος μέλος να μην τους αναγνωρίζονται οι υιοθεσίες. Ε, αυτό το θέμα νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με την λειτουργία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Διότι όταν μετα πα σε ένα άλλο κράτο μέλο και είσαι πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και αποφάσει του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι η ηθαγένεια η ίδια είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχτούν και αστικά δικαιώματα. Και όταν η μη αναγνώριση των δικαιωμάτων του παιδιού ή της υιοθεσία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, τότε είναι βέβαιο ότι αξιοποιώντας τη ρήτρα περί ευρωπαϊκής ηθαγένειας μπορεί να ζητήσουν αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων τα οποία είπατε. Επομένω δεν χρειάζεται μια συνολική ενοποίηση της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, αλλά η αξιοποίηση της ρήτρας της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Και το επόμενο θέμα που πράγματι μας απασχόλησε είναι το ζήτημα των υποχρεωτικών υιοθεσιών. Είδαμε την περίπτωση στη Βρετανία ή στην Γερμανία με το Jugendamt. Τέλος, για τις παρένθετες μητέρες που έθεσε ο συνάδελφος Μαρτάν, τουλάχιστον στην Ελλάδα νομικά το θέμα αυτό έχει αντιμετωπιστεί. Πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε τις διάφορες νομικές πτυχές, αλλά υπάρχουν απαντήσεις νομικές επί του θέματος. Αν υπάρχουν επιμέρους ζητήματα, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τέλο θα κάνω μια ενημέρωση, κυρία Πρόεδρε. Ε, εκ μέρου του ECR ήθελα να σα ενημερώσω. Είμαι μέλο ε, του, του, ε, του Group de Travail, της ομάδας εργασίας για τα θέματα των, του παιδιού. Και αναπληρωματική είναι η κυρία Κάλσον. το ECR λοιπόν σας λέει ότι πλέον τακτικό μέλος στην ομάδα εργασίας θα είναι η κυρία Κάλσον και εγώ θα είμαι αναπληρωματικός. Σας ευχαριστώ να γραφτεί στα πρακτικά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα ε, και καλή επιτυχία με το βιβλίο σας. Ε, okay, let's move on and, ε, Να προχωρήσουμε. Θα εξηγήσω το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει εξή. Υπάρχει μια προθεσμία για τις τροπολογίες στις 3 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 19 Απριλίου και θα περάσει στην Ολομέλεια του Ιουνίου, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη σε όλους όσους ε, εργάζονται επί του πολύ σημαντικού αυτού ζητήματος και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το υπαριθμόν 8. Εγώ τώρα θα πάρω το λόγο να σας μιλήσω για τη γνωμοδότηση για την, έκθεση, την ετήσια έκθεση ε, για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Και η συγγήτρια είμαι εγώ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την Επιτροπή μας και πιστεύω ότι η συνεισφορά μας θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή που είναι βεβαίως η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να μην ξεχνούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη μεταγραφή της νομοθεσίας στην έγκαιρη και την ε, έγκυρη και την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας του ενωσιακού δικαίου στο σύνολό του. Βλέπουμε όμως ε, μέσω των αναφορών που λαμβάνουμε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές περιπτώσεις καθυστερημένης ή κακής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας από καιρού εις καιρών. Πολύ περισσότερα λοιπόν πρέπει να γίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας και ε, ελέγχει κατά πόσο η μεταγραφή της νομοθεσίας συνάδει με τον αρχικό στόχο της νομοθεσίας στο πλαίσιο βέβαια της ε, καλύτερης νομοθεσίας όπως επίσης και ε, της ε, καλύτερης κατάστασης της νομοθεσίας και στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα της νομοθεσίας της Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, όπως είπα και προηγουμένως, πρόκειται για μια γνωμοδότηση και, για, όχι για ένα βιβλίο. Θα ήθελα λοιπόν να σας να είμαστε σύντομοι και ακριβείς και να εστιαστούμε στις ε, αναφορές, τα θέματα των αναφορών που έχουμε λάβει και ελπίζω ότι η συνεισφορά σας θα βελτιώσει το κείμενό μου. Ε, με πολύ χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας ε, για την οριστική εκδοχή του κειμένου μου. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι επίσης η 3η Μαρτίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 19 Απριλίου και θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ε, Ολομέλειας της 23ης Ιουνίου. Θα ήθελε κανείς άλλος συνάδελφος να λάβει το λόγο. Ο κύριος ε, Ζάκη, ε, σκιώδης εισηγητής, δεν είστε υποχρεωμένος, αλλά αν θέλετε να πάρετε το λόγο, πάρα πολύ σύντομα. Σεσίλια, σε γενικές ε, γραμμές, ε, το όραμά σου και οι συστάσει σου είναι, μας βρίσκουν απολύτως ε, σύμφωνους. Κάποιες λεπτομέρειες μόνο θα θέλαμε να ρυθμιστούν με τροπολογίες τις οποίες θα σας υποβάλουμε μέχρι τις 3 Μαρτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Παλ, Εδουάχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι ο εισηγητής του σκιώδους εισηγητή που δεν μπορεί να είναι εδώ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας διαβάσω το, το, σχόλιο της σε σχέση με τη γνωμοδότησή σας. Η συνάδελφη η φως μου λοιπόν να συμφωνεί με τη χρηματοδότησή σας και συμφωνεί και με τους γενικούς στόχους που θέτεται. Είναι μια σωστή οπτική γωνία, δηλαδή να επιμείνουμε στη σημασία των αναφορών που υποβάλλουν ε, οι πολίτες ε, και όπως και η κοινωνία των πολιτών είναι ένας τρόπος να παρακολουθήσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας παρά το γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη το αίτημα της ΠΕΤΗ πέρσι να υπάρξουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας ε, Προ τους αναφέροντες σε σχέση με κοινοποίηση διαφόρων στοιχείων. Ε, η δική σας γνωμοδότηση λαμβάνει υπόψη τη θετική επίδραση του Pilot Project και κάνει μια σημαντική ε, προσπάθεια βελτίωσης όσον αφορά την ενημέρωση για τις εκκρεμείς αναφορές. Η κυρία Μιντι λοιπόν θα ήθελε να δει κάποιες προσθήκες ε, ώστε να συνεισφέρει θετικά στο καλό πνεύμα της γνωμοδότησής σα. Για παράδειγμα, η εφαρμογή συγκεκριμένη και αποτελεσματική ενωσιακή νομοθεσία εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Συνεπώ, πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν ε, να μην επιμένουμε σε μεγαλύτερη, σε πιο μειογενή εφαρμογή τη εφαρμογή, της ε, νομοθεσία τη Ένωση, ε, να υπάρχει ένα μηχανισμό ε, αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών δικτών, όπως επίσης και βάσει συγκριτικής αξιολόγησης και ε, βέλτιστων πρακτικών. Μία πολιτική μηδενικής ανοχής επίσης ενώπιον των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες. Τα κράτη-μέλη σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο και είναι απολύτω σημαντικό να γίνουν σημαντικέ προσπάθειε από πλευρά του ώστε να γίνεται ακριβή εφαρμογή τη νοσιακή νομοθεσία προ όφελο των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης ε, να συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή και μετά τη μεταγραφή της στο εθνικό δίκαιο και να δούμε κατά πόσο στην πράξη γίνεται αυτή, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε διορθωτικούς μηχανισμούς και μηχανικούς αποκατάστασης σε περίπτωση ε, μη ε, ε, εφαρμογή τη νομοθεσία. Η πρόσβαση στην ενημέρωση λοιπόν και η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τις καταγγελίες των πολιτών και όσον αφορά την απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι δικέ μα ερωτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερο στο pilot project του αναφέροντος, να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των πολιτών και των ε, αρμοδίων ε, αρχών όσον αφορά το ΡΕΦΙΤ και την καλύτερη νομοθεσία που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εισηγήτρια για τη δική μας πολιτική ομάδα είναι εξαιρετική σημασία ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, το τα, περιβαλλοντικά θέματα ε, να μην αποδυναμώνονται από όλη τη διαδικασία. Πρέπει τα κριτήρια να είναι σαφή ε, όσον αφορά ε, το άμεσο και το έμεσο, τον, τον άμεσο και τον έμεσο αντίκτυπό τους ε, στην νομοθεσία, όπως επίσης να γίνεται μια ανάλυση της προστιθέμενης αξίας της νομοθεσίας. Η ανάλυση κόστους και ωφέλους πρέπει να συμπεριλάβει κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, διαφορετικά θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι αναφορές των πολιτών κατά τα ερχόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ εκ μέρους της συναδέλφου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη συνάδελφό σας που και τόσο εντατικά. Ήδη από τώρα αποτελεί πολύ μεγάλη πηγή έμπνευσης για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα. Η Ελεονόρα Εύη, θέλετε το λόγο για το θέμα αυτό. Όχι. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Ε, κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με τις ε, βασικές αρχές που διαγράφονται στην γνωμοδότηση την οποία έχετε εισηγηθεί. Ορισμένες παρατηρήσεις θα κάνουμε καταθέτοντας ορισμένες τροπολογίες. Ε, επισημάνω μόνο ότι είναι σημαντική η δραστηριότητα του ελέγχου της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει άμεση σχέση και με την Επιτροπή μας, διότι δεχόμαστε πάρα πολλές αναφορές από τους πολίτες, με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται εδώ και το ότι εμπλέκουμε και την Κομισιόν, λαμβάνει γνώση η Επιτροπή ενδεχομένων παραβιάσεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι η ίδια η διαδικασία της Επιτροπής Αναφορών βοηθά την Επιτροπή, την Κομισιόν, να δει περιπτώσεις παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τις κρίνει και βεβαίως να προχωρήσει ε, σε διαδικασίες που προβλέπουν βλέπονται με βάση τη συνθήκη. Νομίζω βέβαια ότι ε, η απόλυτη διακριτική ευχέρεια που έχει η Επιτροπή, η Κομισιόν στο να προχωρήσει, στο να παραπέμψει ένα κράτος μέλος ή όχι, νομίζω ότι αυτή πρέπει να περιοριστεί κατά την άποψή μας. Δεν μπορεί να είναι απόλυτη διακριτική ευχέρεια, να περνάνε τέσσερα και πέντε χρόνια προκειμένου να γίνουν οι έρευνες και να παραπεμφθεί εδεχόμενα ένα κράτος μέλος για παραβίαση της νομοθεσίας. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το δούμε Παλαιότερα είχα γράψει ένα άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα με παρατηρήσεις διότι πηγάζουν τα ίδια τα δικαιώματα των πολιτών που καταθέτουν τις καταγγελίες είτε μέσω της Επιτροπής Αναφορών είτε απευθείας στην Κομισιόν και δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Κομισιόν να ενεργήσει ή να μην προχωρήσει στην έρευνα και εν συνεχεία στην παραπομπή ενός κράτους μέλους. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και θα κάνουμε παρατηρήσεις με ορισμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για το θέμα αυτό. Ε, υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε το λόγο. Όχι. Ωραία. Να προχωρήσουμε τότε. Πάμε στο επόμενο σημείο. Γνωμοδότηση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής ε, Σύμβασης ε, Ατόμων με Αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τα συμπεράσματα της Επιτροπής UNCRPD. Η συγγήτρια είναι η Ρώσα και της δίνω απευθείας το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταράς. Όπως ε, γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει και προσυπογράφει τη Σύμβαση των ε, Ατόμων με Αναπηρία και φέτος τον Αύγουστο έγινε αναθεώρηση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών της εφαρμογής της συγκεκριμένη σύμβασης από τα κράτη-μέλη εγκρίθηκαν μια σειρά από τελικές παρατηρήσεις, ε, τις οποίες αυτή τη στιγμή συζητάμε. Πρόκειται για συστάσεις ε, τις οποίες έκανε τα Ηνωμένα Έθνη προς ε, όλα τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά για να τηρηθεί η σύμβαση. Εμείς συστήσαμε ένα δίκτυο στο εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συντονιστούμε και να συζητήσουμε αυτές τις παρατηρήσεις. Πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα στην οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Συνήγορος του Πολίτη και ε, ζητήσαμε να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, κρίνει και τι ακριβώς συζητάμε. Ε, εγώ λαμβάνω υπόψη τις συστάσεις 76 και 77 των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ζητήθηκε από την Επιτροπή Αναφορών να συμμετέχει σε αυτό το πλαίσιο. Συζητάμε τώρα κατά πόσον θα πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρμαχος της συμμετοχής μας διότι εμείς δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μένα, αλλά ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εάν συμμετέχει, ε, αρμόδια επιτροπή θα είναι η Επιτροπή Αναφορών, γιατί είναι η μόνη επιτροπή ε, η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και την προάσπιση των συμφερόντων τους, απαντάει στις αναφορές τους και υπερασπίζεται τους ε, πολίτες σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Επομένως, η Επιτροπή Αναφορών μαζί με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή είναι τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι ε, ανεξάρτητα όργανα. Ε, τη γνωμοδότησή μου λοιπόν ε, υπερασπίζομαι την άποψη η Επιτροπή Αναφορών να είναι ε, η αρμόδια για τα θέματα αυτά. Επίσης, Θέλουμε να δεχτούμε τη σύσταση των Ηνωμένων ώστε όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, να την χάνουν εύκολης ε, πρόσβασης, να υπάρχει κείμενα σε μπράιγ, ε, να μπορεί να χρησιμοποιείται η Μπράι στην επικοινωνία με τους αναφέροντες, αυτό γίνεται ήδη και επίσης να μπορεί να χρησιμοποιείται και η νοματική γλώσσα καθώς επίσης και συσκευέ εύκολη ανάγνωσης για διάφορες αναπηρίες αυτής της μορφής. Ε, επίσης έχουμε πολιτικές ε, ένταξης ε, συμβάσεων ώστε να ε, αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού και των υποτροφιών για άτομα με αναπηρία και να λάβουμε υπόψη μας την αναπηρία γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκρίνουμε επίσης τη Διεθνή Μέρα Πρόσβασης της Αναπηρίας το Δεκέμβριο Είχαμε πολύ χρόνο καθυστέρηση, χαιρόμαστε που το συζητάμε το θέμα αυτό. Επίση, αναφέρεται και το θέμα τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία σε όλα τα μέτωπα και επίση αναφερόμαστε και στην εκπαίδευση που περιλαμβάνει του πάντε για να μπορούν όλοι να εντάσσονται στα εκπαιδευτικά συστήματα και να μην υπάρχουν γέτο. Επίση αναφερόμαστε στην κύρωση τη συνθήκη του Μαρακέ για την ε, πρόσβαση όλων των δημοσιευμένων έργων ε, σε άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει συζητήσει επί μακρόν, η Επιτροπή μας έχει συζητηθεί και στην Ολομέλεια, το ε, απασχόλησε και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αλλά αναφερόμαστε σε αυτό γιατί αναφέρθηκε σε αυτό και, ε, αναφέρθηκαν σε αυτό και τα Ηνωμένα Έθνη τον Αύγουστο. Ε, εν είδη συμπεράσματος να σας πω ότι αυτό που κάνει αυτή η γνωμοδότηση ε, δεδομένου ότι θα γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, η Επιτροπή Απασχόλησης ε, και η Επιτροπή των Γυναικών και φυσικά και η Επιτροπή μας. Εγώ είμαι συντάκτρια της γνωμοδότησης και στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Γυναικών. Ξέρετε ότι είμαι και αντιπρόεδρος της ομάδας αρμόδιας για θέματα αναπηρίας και εμείς στο δίκτυο το οποίο δημιουργήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πρικοδότηση από πλευράς γραμματείας ε, για να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά, διότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και οι παρατηρήσει που έγιναν από πλευράς Ηνωμένων Εθνών είναι ε, θέματα τα οποία χρήζουν μελέτης. Ε, ε, είναι προτροπή προς τα κράτη-μέλη για να ε, τηρήσει τα όσα προβλέπει η Σύμβαση και ε, θεωρώ ότι εμείς ως Επιτροπή μπορούμε να έχουμε πολύ ενεργό ρόλο ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι παρατηρήσεις. Μέχρι 3 Μαρτίου οι τροπολογίες, όλες οι παρατηρήσεις λοιπόν που θα κάνετε θα ληφθούν υπόψη και θα ψηφιστεί στις 19 Απριλίου με τις τροποποίησεις που θα έχετε προτείνει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τους κοιόδες εισηγητές. Ε, η Σολεδάδ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ρώσα. Το σχέδιο γνωμοδότησης είναι αρκετά ευρύ. Θα κάνουμε και εμείς τροπολογίες, ε, διότι καλύπτει πολλά ζητήματα. Είναι πολλά τα ευαίσθητα θέματα που θέλουμε και εμείς να σχολιάσουμε. Όπως είπες και εσύ πολύ ωραία, θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν. Για τον τύπο τώρα. Τι θα ζητήσουμε. Βεβαίως τα κράτη-μέλη ε, που δεν το έχουν πράξει ακόμα θα πρέπει να κυρώσουν τη σύμβαση. Ε, είναι πολύ σημαντικό και να υπάρχει και ένας μηχανισμός ελέγχου για να μπορούν τα άτομα με αναπηρίες και οργανώσεις τους να έρχονται σε επαφή και να υπάρχει μόνιμη παρακολούθηση για τα δικαιώματα των παιδιών, των ανθρώπων αυτών. Συγγνώμη. Επίσης, θέλουμε να επιμείνουμε στα εξή θέματα. Τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται ειδική μνήμα στα παιδιά. Πολύ νωρί να υπάρχει ποιοτική εκπαίδευση με συμμετοχή των παιδιών σε όλη τη διαδικασία. Από τους αναπήρους γενικά τα παιδιά με αναπηρίες είναι εκείνα που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες να πούν τι προβλήματα έχουν, τι ανάγκες και θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός που να τα βοηθάει και να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και να μιλούν για τις αγωνίες, τους φόβους τους κτλ. Και νομοθετικά να καλύπτεται. Γυναίκες επίσης με αναπηρία. Θα πρέπει να υπάρχει και μια διάσταση φύλου. Ξέρουμε ότι η ανάπηρη γυναίκα έχει διπλή διάκριση να αντιμετωπίσει. Και για την απειρία και για το γεγονός ότι είναι γυναίκα. Οπότε θα πρέπει να είναι αυτόνομοι και οι άνθρωποι με τις αναπηρίες. Και άλλο σημαντικό στοιχείο να δούμε τι δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν. Υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία ε, να είναι αυτόνομοι οι άνθρωποι αυτοί και να μπορούν να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα να προβαίνουν σε ε, τέτοιες πράξεις και να είναι απολύτως αυτόνομοι και αυτοεξυπηρετούμενοι. Ακόμα και για να ψηφίσει κανείς, ξέρετε, σε πολλές χώρες υπάρχει στενή ερμηνεία ε, της δυνατότητας να δράσει κάποιος και τον έχουν υποκειδαιμονία και δεν μπορεί να διαχειριστεί την ίδια του τη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουν πρόσβαση και στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι με αναπηρίες, έχουν οικονομικές δυσκολίες, δυσκολίες εργασιακές, ε, δεν έχουν ε, υψηλή αγοραστική δύναμη και η δικαιοσύνη θα πρέπει να τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Όταν πρόκειται για θέματα αναπηρίας θα πρέπει να είναι εγγυημένη και να μην υπάρχει κανένα είδους εμπόδιο. Η δικαιοσύνη να είναι τελείως δωρεάν και καθολική η κάλυψη. Επίσης θα πρέπει να γίνει λόγος για την οικογένεια για τους ανθρώπους που είναι το περιβάλλον των αναπήρων, τους υποστηρίζουν και τους βοηθούν. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα άτομα με αναπηρία. Ξέρετε ότι χρειάζεται μια ολόκληρη οικογένεια για να στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα ανάλογα με εκείνους που έχουν τα περισσότερα, μεγαλύτερα ποσοστά αναπηρία. Και να ξεκινήσουν τα διάφορα προγράμματα από τα θεσμικά όργανα για να μπορούν οι άνθρωποι να βοηθούν ε, τους αναπήρους τους. Και για την υγεία δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις εκεί στην πρόσβαση των ε, υπηρεσιών υγείας, δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Πολλές φορές θεωρούμε ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν λιγότερα δικαιώματα ή λιγότερες ε, ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το θέμα της συνένεσης κατόπιν ενημέρωσης και για ζητήματα υγείας ε, για να μπορούν ε, άνθρωποι να παίρνουν τις αποφάσεις τους και επίσης να γίνεται λόγος για κέντρα αναφοράς που ασχολούνται με την αναπηρία. Και ένα τελευταίο, να μιλήσουμε και για ευρωπαϊκό χώρο πρόσβασης ή προσβασιμότητας. Υπάρχει σχετική έκθεση γνωμοδότηση της κυρίας Εσταράς. Θα πρέπει όμως, το ανέφερε προηγουμένως και η συγκήτρια, να γίνεται λόγος για ένα ευρωπαϊκό χώρο προσβασιμότητα και εδώ δεν μιλάω για φυσικά εμπόδια να έχουν πρόσβαση φυσική αλλά στα κοινωνικά δικαιώματα και στα γενικότερα δικαιώματα. Να υπάρχει μια εναρμονισμένη ενημέρωση δεν λέμε στο κάθε κράτο μέρο πώς θα πρέπει να χειρίζεται τα αυτά τα θέματα, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίσουν όπως στην ιατρική υπάρχουν διεθνεί ταξινομήσεις και ξέρουμε τι η κάθε ασθένεια, κάπως θα πρέπει να εναρμονίσουμε τη διάγνωση για την εκάστοτε αναπηρία και πώ απονέμεται το, το μάλλον, πώς ταξινομούνται οι ανάπηροι ανάλογα με την αναπηρία τους. Επίσης, η ψηφιακή ατζέντα. Μιλάμε για μια ψηφιακή εποχή. Είναι κρίμα να μην γίνεται κανένα λόγο στο θέμα αυτό και στην έκθεση για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. It's... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό να έχουμε συναδέλφους ε, που πραγματικά συμμετέχουν στη συζήτηση, όμως ε, είναι μια γνωμοδότηση, μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε όλα τα σχετικά θέματα, απλώ και μόνο τα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Εκ μέρου των φιλελευθέρων, ε, σκιώδη συγγήτρια η Μπεατρής, έχουμε 40 λεπτά χάσει. Και μετά ο κύριος Μαριάς. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα στο που θα εστιάσουμε. Ε, συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση της κυρίας Εσταράς και να πω ότι αυτό που έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι να διαθέτουμε ένα σημαντικό μέσο όπως είναι αυτή η διοργανική ομάδα για την αναπηρία και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά προς αυτή την κατεύθυνση με βάση αυτό και επίσης να λάβουμε υπόψη μας και την ε, ε, περίοδο τη μεταβατική διαβουλώσεως που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η γνωμοδότησή μας πρέπει να έχει κάποια προστιθόμενη αξία και αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε που ήσουν τόσο σύντομη, Μπεατρή. Αυτό είναι καλό παράδειγμα. Ο κύριος Μαριάς, ελπίζω να ακολουθήσετε κι εσείς το παράδειγμα. Να ε, πω ότι συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση της κυρίας Σεσταρά ε, ήδη έχουμε κάνει και συζητήσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, έχουμε κάνει και κάποια εκδήλωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ε, ε, σύμβασης ε, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ ε, και επίσης πρέπει να προχωρήσουμε και στην ε, κύρωση της συνθήκης του Μαρακές. Νομίζω ότι τα θέματα που φύγονται είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να υπάρξει στήριξη των ατόμων με αναπηρία, ιδίως σε μια φάση τεράστιας οικονομικής κρίσης, ε, συνολικά στην Ευρώπη, αλλά ειδικότερα και σε χώρες οι οποίες πλήττονται από το μνημόνιο, όπως είναι η Ελλάδα, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσβασιμότητας στα άτομα με ειδικέ ανάγκες και στην υγεία και στα φάρμακα και στην απασχόληση και σε όλες τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να μας απασχολήσει. Τα υπόλοιπα θα τα επισημάνουμε και με ενδεχόμενες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ελεονόρα. Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ πολύ σύντομα. Ήθελα απλώς ε, να πω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα στη γνωμοδότηση αυτή. Είναι η περιβαίωτη μετάβαση από την ε, θεραπεία ε, στα, νοσοκομεία και στα Ινστιτούτα ε, σε μια θεραπεία που βασίζεται στην οικογένεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και εναρμόνιση των δικαιωμάτων των ατόμων που φροντίζουν άτομα με αναπηρία ή και με βαριά αναπηρία. Διότι το πρόβλημα είναι ότι σε πολλέ χώρε, όπω και στην Ιταλία, δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα σε αυτού του ανθρώπου. Επομένω, θα θέλαμε και εμεί ε, να προτείνουμε να ληφθεί και αυτή η πτυχή υπόψη. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλπιόλ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί θα κάνουμε και εμεί τροπολογίε όταν έρθει η ώρα του. Αλλά θέλαμε να επιμείνουμε σε δύο θέματα. Πρώτον, την ανάγκη να υπάρχουν δημόσιοι πόροι, γιατί οι κυβερνήσει θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ζωή για όλου του ανθρώπου και για τα άτομα με αναπηρίε. Είδαμε τα τελευταία χρόνια τι έγινε. Ακριβώ με τι πολιτικέ των μνημονίων και τη λιτότητα κλείσανε ειδικά κέντρα, ε, ειδικά ε, εργαστήρια, θέσει απασχόληση. Τα κόψαν όλα αυτά τα μνημόνια και μετά είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στην πολιτική συμμετοχή στη δημόσια ζωή των αναπήρων. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία στο άρθρο 29 λέγει ότι τα κράτη εγγυώνται το δικαίωμα των προσώπων αυτών να συμμετέχουν στην πολιτική, στην κοινωνική ζωή, στη δημόσια ζωή. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται το δικαίωμα αυτό και στο Ισπανικό κράτος είναι 80.000, 80.000 παρακαλώ, που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές, διότι τους θεωρούν ανίκανους ε, ε, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις σχετικές. Ε, ο ΙΕ έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στο Ισπανικό κράτος για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, πράγμα που δεν έπραξε το κράτος της Ισπανίας θα το θέσουμε αυτό και ε, θα το ζητήσουμε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την Ισπανία, γιατί οι άνθρωποι έχουν δημοκρατικά, πολιτικά δικαιώματα και ατομικά και δικαίωμα συμμετοχή στα κοινά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο. Please go ahead. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σύντομα. Καταρχάς να σας πω ότι αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης μας φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μάθω κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να υπάρχει ένα σημείο 11 λίγο σαφέστερο όσον αφορά το τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον ακριβέστερο ορισμό ε, της αναπηρίας, δεδομένου ότι υπάρχει ορισμός αυτό στη σύμβαση. Θα θέλα λοιπόν λίγες περισσότερες εξηγήσεις. Και επίση να σα ενημερώσω για το εξή, ότι βεβαίω συμφωνούμε με την κύρωση του επιπρόσθετου πρωτοκόλλου, αλλά υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που τίθενται. Η γνωμοδότηση ακριβώς αναφέρει ότι πρέπει να αποσαφινιστούν ε, πριν προχωρήσουμε για να μην υπάρξουν εκπλήξεις όπως υπήρξαν με το μηχανισμό επίβλεψης θα επανέλθουμε λοιπόν στο Κοινοβούλιο ε, ως προς αυτό και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας ε, όσον αφορά το European Accessibility Act, το οποίο βεβαίως θα συζητηθεί και στη δική σας Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η Ρώσα μας είπε ότι δεν θέλει να λάβει το λόγο ξανά. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 3 Μαρτίου, 19 Απριλίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και κατά πάσα πιθανότητα ε, θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη Ολομέλειας του Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην συνεδρίαση των συντονιστών, οπότε θα ήθελα να ζητήσω από όλους όσους δεν δικαιούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση των συντονιστών ε, να αποχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.